Σας παρακαλώ, θα ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης. Μας τιμά η παρουσία της εξοχότητάς του. Ταμπού Μομπέκη, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτιού Αφρικής και Προέδρου της του πάνελ υψηλού επίπεδου για την εφαρμογή των μέτρων για το Σουδάν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Μπέκη για τον ενδιαφέρον που έδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ενδιαφέρον του να συναντηθεί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κοινή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξη. Αργότερα πρόεδρος Μπέκη θα συναντηθεί με την, Επιτροπή, την Πολιτική Επιτροπή και την Πολιτική Ασφάλειας. Μετά θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, τη Λέδη Άστον. Ο πρόεδρος Μπέκη συνοδεύεται από την εξοχότητά του Πιέρ Μπουγιόια, πρώην πρόεδρο του Μπουρούντι. Τον χαιρετίζουμε ο οποίος είναι μαζί μας εδώ στο βήμα και από τον πρέσβη Μοχάμπεντα Λαντίφ που επίσης ε, καλωσορίζω θερμά. Θα θέλαμε να συζητήσουμε την κατάσταση στο Σουδάν και τις επικείμενες εκλογές εκεί που είναι σημαντικές και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν ερωτήσεις να υποβάλουν και θα σας παρακαλούσαμε να πάρετε το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή επί του θέματος. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πραγματικά που μας διαθέτετε κάποιο χρόνο να είμαστε εδώ μαζί σας να συζητήσουμε ένα θέμα που ανέφερε ο πρόεδρος μας εδώ, το Σουδάν δηλαδή. Όπως προανέφερε, ανήκουμε στην Αφρικανική Ένωση, στην ομάδα υψηλού επίπεδου της Αφρικανικής Ένωσης για την εφαρμογή στο Σουδάν του σχεδίου. Τέλος Οκτωβρίου δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, πέρσι, και εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή της Αφρικανικής Ενώσης, το πάνελ, στην ομάδα μας είναι να βοηθούμε, να βοηθήσουμε το Σουδάν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από την ηρευτική Συμφωνία που συνήθει μεταξύ Βορρά και Νότου υπεγράφει το 2005 όπως τα ξέρουν τα μέλη του Κοινοβουλίου και άλλα συναφή θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να λυθεί το, η σύγκρουση στο Νταρφούρ και να βοηθήσουμε το Σουδάν όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και εκλογές που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 11 Απριλίου. Αυτή είναι η εντολή που μας δόθηκε. Εν γέννη, λέω σε όλους, ότι θα πρέπει να προσέξουμε ό,τι κινείται στο Σουδάν, ό,τι γίνεται στο Σουδάν. Τι κάνει λοιπόν αυτό το πάνελ, αυτή η ομάδα, προσπαθεί να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις στο Σουδάν, και να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις και πρέπει να σας πω βεβαίως κάτι που θα γνωρίζουν τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι για την Αφρικανική Ήπειρο το Σουδάν έχει ιδιαίτερη θέση στην Ήπειρό μας. Είναι πολύ μεγάλη χώρα. Έχει κοινά σύνορα με άλλες 9 Αφρικανικές χώρες και είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι αν κάτι πάει πολύ στραβά, πολύ άσχημα στο Σουδάν, θα επηρεάσει όχι μόνο τη γειτονική περιοχή αλλά την Ήπειρο στο σύνολό της. Οπότε η επίλυση των προβλημάτων του Σουδάν ε, γίνεται πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και γι' αυτό η Αφρικανική Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την ομάδα, αυτό το πάνελ, με μια συγκεκριμένη εντολή με πολλά θέματα, ούτω ώστε η Ήπειρος να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και των συγκρούσεων. Οι εκλογές έρχονται, έχουν προγραμματιστεί για τις 11 Απριλίου, είναι περίπλοκο ζήτημα, είναι περίπλοκες ε, εκλογές, πρέπει να ψηφιστεί πρόεδρος, κοινοβούλιο, τοπικό, περιφερειακές εκλογές, αλλά δυστυχώς από τούδε και στο εξή όλες οι πολιτικές δυνάμεις στο Σουδάν ευτυχώ συμμετέχουν στις εκλογές παρά τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν όλοι όμως θέλουν να συμμετάσχουν στι εκλογές και σαν πάνελ προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε όλους να παραμείνουν εντός της εκλογικής διαδικασίας. Γιατί το λέω αυτό, διότι υπήρχαν πολλές απειλές, πολλοί απειλούσαν θα αποσυρθούν από τις εκλογές εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι, να παραμείνουν όλοι και τα προβλήματα, τα ιαδήποτε προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν. Σαν πάνελ προσέχουμε αυτά τα ζητήματα, θέλουμε να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς και η ε, Επιτροπή των Εκλογών και να επιληθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και να υπάρχουν επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα ούτω ώστε να παραμείνουν τα πολιτικά κόμματα εντό εκλογική διαδικασία. Σαν τμήμα τη προσπαθία αυτή, κατόπιν αιτήματο των πολιτικών κομμάτων, συντάξαμε ένα διοντολογικό κώδικα με τον οποίο συμμορφώνονται όλοι εθελοντικά. Θα συμμορφώνονται τα κόμματα εθελοντικά, όλα τα μέρη τα εμπλεκόμενα και δημιουργήθηκε ομάδα εποπτική στο Σουδάν η οποία θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει την εφαρμογή του εν λόγω διοντολογικού κώδικα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών. Αυτή την προσπάθεια έχουμε ξεκινήσει και είναι σημαντικό το, το κομμάτι της όλης διαδικασίας των αλλαγών στο Σουδάν, διότι το πάνελ πιστεύει επίσης ότι αν το κλίμα και η ατμόσφαιρα και οι συνθήκες δημιουργηθούν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Σουδάν, τότε η διαδικασία του εκδημοκρατισμού της χώρας ε, θα προχωρήσει και είναι κάτι που έχει κρίσιμη σημασία. Είναι το θέμα του Νταρφούρ βέβαια μετά. Διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις στην Τόχα, στο Κατάρ και ουσιαστικά είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ των ε, αντιμαχόμενων πλευρών, ενόπλων. Δηλαδή κυβέρνηση από τη μια μεριά, επαναστατικές ομάδες από την άλλη. Ε, βασικό στοιχείο είναι η προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός και άλλα συναφή θέματα για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτή η διαδικασία ε, προχωρά πιο πέρα θέλουμε να επιτευχθεί μια γενική πολιτική συμφωνία. Γίνονται οι πραγματεύσεις και με αυτό το σκοπό, δοθέντος του τι συμβαίνει τώρα και της προσοχής που δίδεται στις εκλογές, νομίζω ότι οι γενικές διαπραγματεύσεις που θέλαν να πετύχουν μια γενική πολιτική συμφωνία πιθανότατα να λάβουν χώρα από τη στιγμή που θα λήξουν οι εκλογές και θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση αλλά η πρόοδος ε, που έχει σημειωθεί τώρα με την υπογραφή των εγγράφων για την κατάπαυση του πυρός είναι βέβαια πολύ σημαντική. Αλλά επίσης ε, πολύ σημαντική είναι για, την για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει σε μια πιο καθολική πολιτική συμφωνία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο όσους συμμετέχουν στις εκτροπραξίες, αλλά θα πρέπει να διευθετείται και το θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων μας είπαν οι άνθρωποι αυτοί ότι θέλουν να εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις. Ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που θίγονται από τη σύρουξη αυτή και θα πρέπει να μπορέσουν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν ε, σε αυτή την... έχουμε αυτή τη διαδικασία τη συμμετοχική που θα πρέπει να λάβει χώρα. Γενικά ε, μεταξύ των κατοίκων του Δερφούν υπάρχει συμφωνία, έχουμε το θέμα του καταμερισμού, της πολιτικής εξουσίας ε, και άλλων θεμάτων, αναπτυξιακών θεμάτων κτλ. Και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη συμφιλίωση. Συζητείτε το θέμα αυτό, το συζητά το πάνελ με την κυβέρνηση του Σουδάν έτσι ώστε όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή να γίνουν αυτές ε, οι καθολικές διαπραγματεύσεις και όλοι να είναι σε θέση να μπορούν να λάβουν αποφάσεις για το πώς θα προσεγγιστεί το θέμα της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης, γιατί όλοι συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια της σύραξης στον Τερφούρ ε, έγιναν ε, πολλά εγκλήματα, και επομένως στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και το ερώτημα <laughs> είναι πώς αποδίδεται η δικαιοσύνη αυτή. Έτσι λοιπόν, εδώ σας δηλώνω ότι κάναμε κάποιες ε, προτάσεις ε, για το θέμα αυτό, θα το γνωρίζετε. Και ε, φυσικά θέλουμε να δεσμεύσουμε και την κυβέρνηση του Σουδάν επί του θέματος αυτού, έτσι ώστε τη στιγμή που θα λάβουν χώρα αυτές οι καθολικές διαπραγματεύσεις να είναι δυνατόν να επιληθούν τέτοια ζητήματα. Επομένως, ε, θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση ως προς την ανάληψη δεσμεύσεων για τις συνολικές διαπραγματεύσεις, ε, τις καθολικές διαπραγματεύσεις του Νταρφούρ λόγω των επικείμενων εκλογών, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία εξελίσσεται όπως και να έχει. Φυσικά το δημοψήφισμα στο οποίο θα συμμετάχουν οι πολίτες του Σουδάν για να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν εντός του Σουδάν ή όχι. Θα γίνει του χρόνου τον Ιανουάριο. Και όταν αναλάβει η χώρα αυτό το δημοψήφισμα, θα πρέπει να γίνει υπό μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν χώρα οι εκλογές για να υπάρχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση όταν θα λάβει χώρα και το δημοψήφισμα και θα αποφασίσουν οι πολίτες αν το Νότιο Σουδάν θα παραμείνει πτήμα του Σουδάν ή αν θα αποσχιστεί. Η συνέπεια φυσικά είναι ότι υπάρχει αναγκαιότητα να δούμε τα θέματα μετά το δημοψήφισμα. Δηλαδή, αν το Νότιο Σουδάν ψηφίσει υπέρ της ανεξαρτησίας, τι θα γίνει με το θέμα των πολιτών, με την περιουσία, με το πετρέλαιο, όλα αυτά τα πράγματα. Παρόμοια ερωτήματα προκύπτουν ε, για το τι θα γίνει αν ψηφίσει ο πληθυσμό για ένα ενωμένο Σουδάν. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι η ενότητα ε, θα υλοποιηθεί ουσιαστικά υπό το σημερινό καθεστώς, υπό τις σημερινές διευθετήσεις, ακόμη και αν αποφασίσουν να διατηρήσουν τη χώρα ενωμένη. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Υπάρχουν προετοιμασίες για το θέμα αυτό, για να λυθούν τα θέματα μετά το δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους ή νωρίτερα. Γιατί τη στιγμή που θα πάνε να ψηφίσουν στις 9 Ιανουαρίου 2011 οι πολίτες θα πρέπει να υπάρχουν ε, αυτές οι επιλογές. Έτσι λοιπόν οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα κατόπιν του ψηφίσματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και θα πρέπει ουσιαστικά να συμπεριληφθούν στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα έτσι ώστε κάποιος ε, που θα πάει να ψηφίσει να μπορεί να κάνει μια επιλογή κατόπιν ενημέρωσης. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να σταματήσω για το θέμα αυτό, όπως μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, υπάρχουν ε, πολλά επίγοντα θέματα, σημαντικά αλλά και επίγοντα που θα πρέπει να επιλύσουμε. Και επειδή μας πίζει ο χρόνος, είναι δύσκολο να πούμε ε, με αυτή την προτεραιότητα ασχοληθούμε τη Δευτέρα και με την άλλη την Παρασκευή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες και να πω ότι εν τέλει ελπίζουμε ότι τελικά θα υπάρξει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση που θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος του Ντερφούρ μέσα στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού του Σουδάν και θα επιλύσει το θέμα της σύραξης έτσι λοιπόν ακόμη και αν οι πολίτε του Νότιου Σουδάν ψηφίσουν υπέρ τη ανεξαρτησία. τότε το θέμα των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών είναι αντικείμενο διαχείριση. μιας φιλικής διαχείρισης. Παρά μιας διαχείρισης που θα προκαλεί τριβές. Γιατί Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί δεσμοί μεταξύ Βορρά και Νότου. Επομένω, ε, θα πρέπει να εξεύρουν έναν τρόπο αρμονική συμβίωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ ενημερωτικά τα όσα μας είπατε και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από το φίλο και συνάδελφο από την ε, Επιτροπή Ανάπτυξη τον κύριο Ντέβα να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πραγματικά μας ε, παρουσιάσετε κάποιες ε, πολύ θερμές προσδοκίες για το μέλλον του Σουδάν και μάλλον μόνο εσείς και ε, πολύ λίγοι θα μπορούσαν να, να μας αναφέρουν να μας παρουσιάσουν τέτοια αποτελέσματα, γιατί είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτό περί συμφιλίωσης που μας παρουσιάσατε σε σχέση με το Σουδάν. Και στο πλαίσιο αυτό ήθελα να σας ενημερώσω ότι αργότερα σήμερα η Επιτροπή αυτή και η δική μου Επιτροπή θα συζητήσουν ε, με τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο οποίος, ε, τον, οποίο το έργο υποστηρίζουμε τα μάλα. Κατά την άποψή σας, ε, τι θα έπρεπε να πούμε στον επικεφαλής εισαγγελέα. Δεύτερον, και σας ρωτώ φιλικά. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο να λάβει κάποιο δράσει για να προλάβει τραγωδίε που βλέπουμε να εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μα στην Αφρική. Πού είναι η έννοια της πρόληψης, ε, της ανάληψης δράσης εκ των προτέρων. Δεν ε, απευθύνω βέβαια σε εσά ε, ακριβώ την ερώτηση αυτή. Δεν πει να ρωτήσω, αλλά γιατί πρέπει τελικά τόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι να υποφέρουν ε, και να πεθάνουν πριν να κάνουμε κάτι. Έχουμε εδώ και τον πρόεδρο του Μπουρουντή και απευθύνομαι και σε αυτόν. Γιατί χρειάζεται τόσο, τόσο πολύ καιρό για να σώσουμε ζωές. Ναι, αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Κυρία Ντεκάιζερ, παρακαλώ. Είναι επικεφαλής ε, παρατητής ε, της ε, Ευρωπαϊκής Αποστολής Παρακολούθησης των Εκλογών στο Σουδάν, Βερόνικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους Προέδρους, μάλλον. Και ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την δράση που αναλαμβάνετε πέρσι της Ειρήνης και κυρίως ευχαριστώ τον κύριο Μπέκη Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές ε, όχι μόνο θα γίνουν τον Απρίλιο, κάτι που φαίνεται σχεδόν βέβαιο σήμερα, αλλά ελπίζω να υλοποιηθούν ε, με ένα τέτοιο τρόπο που θα ανοίξουν το δρόμο για την ειρήνευση στο Σουδάν. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει μια τόσο μεγάλη αποστολή για να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι υποστηρίζει και θα υποστηρίξει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Τώρα, Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε συζήτηση ούτε για τη μερομηνία των εκλογών, ούτε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ξέρουμε, όλα σου έχουν υποθεί για το θέμα αυτό. Αλλά να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας και στη διαδικασία την ειρηνευτική. Δεν μιλάω για το ρόλο των κρατών μελών, αλλά βλέπετε να υπάρχει εδώ ρόλος να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μέχρι τώρα τελικά μάλλον ήταν κάπως απούσα, έχει φανεί κάπως απούσα. Μήπως ε, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένας πιθανός ρόλος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία, τη μετακλογική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες, που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για την επιτήρηση των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκλογές του Σουδάν, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει μικροφόνο μικροφώνου κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε Εμπέκη για την παρουσίασή σας. Δεν θα μακρηγορήσω επί των θεμάτων που αναφέρατε όπως τα θέματα ε, δικαι... απόδοσης δικαιοσύνης του Νταρφούρ και το μέλλον του Σουδάν. Ε, αναμονή το αποτελεσμά της συμφωνίας Νεβάσα αλλά θέλουμε να εστιαστούμε επί της προετοιμασίας των εκλογών. Εξεπλάγει από μια δήλωση που διάβασα του Προέδρου Αμπασίρ στα μέσα ενημέρωση που διατείνεται ότι θα κόψετε τα δάχτυλα των παρατηρητών και όταν συνθλίψετε τους παρατηρητές θα τους συντρίψετε. Αυτή είναι η αντίδραση όσον αφορά αυτά που είπε το κέντρο Κάρτερ ότι θα καθυστερήσουν οι εκλογές λόγω των, της προετοιμασίας. Ποια είναι η άποψη σας, η δική σας ή του Πρόεδρου Μπούγια θα μπορούν να συμμετέχουν εσωτερικοί παρατηρητές πέραν των διεθνών παρατηρητών, θα τους επιτραπεί να κάνουν τη δουλειά τους. Η, η αρμόδια επιτροπή της εκλογές μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανεξαρτησία της για να επιλύσει ενδεχόμενα προβλήματα. Θα υπάρχει ελευθεροτυπία, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Κάτι κρίσιμο για την εκλογική διαδικασία. και είστε ικανοποιημένος όσον αφορά τις συνθήκες που θα επικρατούν για τη σωστή καταμέτρηση των ψήφων. Αυτό είναι απαραίτητο για τις εκλογές. Είδαμε σε πολλά μέρη ότι παρόλο που όλα πάνε καλά μέχρι την ημέρα των εκλογών όσον αφορά την καταμέτρηση των ψήφων τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Αν μπορείτε, μπορείτε να εκφράσετε κάποιες απόψεις πάνω σε αυτό. Εάν θεωρείτε βέβαια ότι είναι φρόνιμο να εκφράσετε απόψεις επ' αυτών. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες, λέει ο Πρόεδρος. Καλό τον κύριο Μπέκη, τον πρόεδρο Μπέκη, να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων και να πούμε σε όλους ότι υπάρχουν άλλοι τέσσερις συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Θα ακουστούν όμως αφού δώσετε εσείς κύριε Πρόεδρε πρώτα τις ε, απαντήσεις σας. Έχετε το λόγο. Όσον αφορά το, τον εισαγγελέα και την δίωξη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ήρθαμε σε επαφή με τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όσον αφορά τα θέματα δικαιοσύνης και τα θέματα που απορρέουν από το πρόβλημα του Νταρφούρ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Μας είπε ότι πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ε, τε, τελεσίδικο δικαστήριο, δηλαδή ε, δρά συμπληρωματικά σε σχέση με, το, με τα εσωτερικά δικαστικά συστήματα των χωρών. Και το δικαστήριο εξέδωσε διάφορα εντάλματα όσον αφορά το Σουδάν, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, τα εντάλματα αυτά, να θεωρηθούμε ότι είναι κάτι δοθέν, είναι δεδομένο. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό θα είναι να κάνει τους δικαστές του δικαστηρίου να αλλάξουν γνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι δεδομένο μας είπε, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αντιμετωπίσει όλα τα εγκλήματα που ενδεχομένως έχουν διαπραχθεί στο Νταρφούρ. Και γι' αυτό θα είναι σημαντικό η Επιτροπή μας, το πάνελ μας, να εξετάσει τι μπορεί να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει εσωτερικά, εντός Σουδάν, για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα εγκλήματα, να εξηχνιαστούν. Και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, δεν θα ήθελε να αντικαταστήσει οδήποτε εσωτερικό δικαστικό σύστημα χώρας. Και όσον αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν το Σουδάν και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είχαν καμία πρόθεση να ε, απαγγείλουν κατηγορίες κάτι οδήποτε και να απαγγείλουν, να εκδώσουν και άλλα εντάλματα. Το βάρος ουσιαστικά είναι στο εσωτερικό δικαστικό σύστημα της χώρας. Το συζητήσαμε λοιπόν το θέμα σε αυτό το πλαίσιο ε, και κάναμε διάφορες προτάσεις όσον αφορά τη συμφιλίωση και τη δικαιοσύνη συμπεριλάβαμε και κάποιες προτάσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμό του Νταρφούρ που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην εξαρτησία του δικαστικού συστήματος του Σουδάν και κάναμε προτάσεις πώς μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη στα θύματα των διαπραχθέντων εγκλημάτων. Εξού και η ιδέα του υβριδικού δικαστηρίου κλπ. Να φέρουμε και εξωτερικούς δικαστές, ερευνητές, εισαγγελείς από το εξωτερικό να έρθουν στο Σουδάν και να βοηθήσουν τις έρευνες, τη δίωξη και την εξυχνίαση των διαφόρων υποθέσεων και την εκδίκασή τους. Ο κ. Σοκάμπου ε, είμαι σίγουρος ότι θα σας πει παρόμοια πράγματα όσον αφορά το Σουδάν. Δεν χρειάζεται να, να, του πείτε τίποτα για το Σουδάν. Αυτά θα πει, αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει τέλεια συνεννόηση μεταξύ του πάνελ και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της δικαιοσύνης. Και αυτή την αντιμετώπιση την δέχονται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ας πέρασουμε τώρα στις άλλες ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά είναι πολύ σημαντικός εταίρος της Αφρικανικής Ένωσης σε πάρα πολλά ζητήματα και συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της ειρήνης και της ε, επίλυσης των συγκρούσεων. Αυτό θα πρέπει, αυτή η συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν, τον πρεσβευτή Πράιλ. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Συναντηθήσαμε ε, σήμερα το πρωί τον Επίτροπο ανάπτυξη και του είπαμε ότι εμεί ω πάνελ θα ζητήσουμε κάποια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το πάνελ θα πρέπει να αναπτύξει και τη δική του ικανότητα να μπορέσει να παρέχει συμβουλέ για διάφορα προβλήματα είτε αφορούν το πετρέλαιο, είτε αφορούν τα σύνορα. Και χρειαζόμαστε εμείς λοιπόν ως πάνελ υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποκτήσουμε αρμοδιότητα για να κάνουμε κάποιες συμβουλές και κάποιες ε, προτάσεις. Δηλαδή όχι ε, να βγάζουμε από το κεφάλι μας ε, διάφορες προτάσεις, αλλά να μπορούμε να έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Αν δούμε τώρα το θέμα του Νταρφούρ, ένα από τα ουσιαστικά θέματα για την επίλυση της σύραξης είναι το αναπτυξιακό ζήτημα και αυτό το θέτει και ο πληθυσμός πρέπει να δούμε πώς αναπτύχθηκε το Σουδάν ιστορικά σε μια μεγάλη χρονική περίοδο και επειδή αναπτύχθηκε κατά συγκεκριμένο τρόπο και επειδή μια μειονότητα είχε το μονοπόλιο της εξουσίας, το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ουσιαστικά απομόνωση, περιθωριοποίηση των διάφορων περιφερειών και του Νταρφούρ. Και αν θέλουμε να επιλύσουμε τη σύραξη στο Νταρφούρ, πρέπει να αποκατασταθεί και η ισορροπία. Πρέπει να διορθωθούν τα προβλήματα που είχαν τεθεί στο παρελθόν. Και αυτό αφορά και το θέμα της ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, ε, τον Επίτροπο συζητήσαμε το θέμα των περιφερειών. Ε, αυτό το θέμα του Νταρφούρ ε, ουσιαστικά είναι το ίδιο. Αφορά τον Νότιο Σουδάν. Έτσι λοιπόν, η δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα, στον τομέα αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ακόμη και αν ε, τελικά καταλήξουμε στο να έχουμε δύο χώρε πάλι θα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη και αν παραμείνει ενωμένη χώρα, εξακολουθούν να παραμένουν οι προκλήσεις. Η Αφρικανική Ένωση φυσικά και θα ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διερευνήσει τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν όπως ε, σας είπα, επειδή είναι τόσο σημαντική η χώρα αυτή για την Αφρικανική Ήπειρο, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να μεταμορφώσουμε το Σουδάν σε ένα παράγοντα σταθερότητας για την Ήπειρο. Πιστεύω ότι οι Αφρικανοί προσπαθούν να, να σταματήσουν νωρίς, εγκαίρως τις σειράξεις. Αυτό αληθεύει. Αλλά να σας πω ότι βάσει της δικής μου εμπειρίας Ούτως ή άλλως η πυλή των σειράξεων παντού στον κόσμο είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ένα από τα προβλήματα που υπάρχει σε κάθε σύραξη σχεδόν είναι ότι κάθε πλευρά έχει δίκιο. Θα θυμάστε, λόγου χάρη, στη σύραξη στην ακτή του Αλεφαντεστού... Είχαμε τους ε, επαναστάτες οι οποίοι κατέλαβαν το βορείτημα της χώρας και έτσι διέρεσαν τη χώρα στα δύο. Εμείς προσπαθήσαμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Πήγαμε, συζητήσαμε με τον πρόεδρο ε, και είπαμε ωραία δίκιο έχετε και συζητήσαμε και τον Αμσόρου και ε, ουσιαστικά και αυτοί είχαν το δίκιο τους. Επομένως, τελικά πρέπει να συζητήσει κανείς και με τα δύο μέρη και να πει «Ωραία, και οι δύο έχετε το δίκιο σας. Πώς ε, τώρα θα επιλύσουμε όμως το πρόβλημα και θα καλύψουμε τα αιτήματα» όλων των πλευρών. Χρειάζεται χρόνος. Δεν υπάρχει λοιπόν πουθενά στον κόσμο επίλυση, δυνατή επίλυση μιας κρίσης με το να επιβάλλουμε λύσεις. Πουθενά, ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στο Κασμίρ, στο Κονγκό, στο Σουδάν. Χρειάζεται χρόνος για την επίλυση των σειράξεων, όχι γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να δράσουν. Η Αφρικανική Ένωση προσπάθησε να αναπτύξει αυτό που λέμε early warning capacity, ικανότητα έγκαιρη προειδοποίηση, προκειμένου να μπορούμε να ανοιχνεύουμε έγκαιρα θέματα που θα οδηγήσουν σε προβλήματα. Όμως φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αν έρθετε σε μένα ως ε, πρόεδρο της ε, Νοτιομουφρικής και μου πείτε ε, σε δύο χρόνια θα ξεσπάσει σύγκρουση, εγώ θα πω, α, πώς το ξέρεις, δική μου είναι η χώρα. Όμως ε, το θέμα είναι ότι με αυτό το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να μπορούμε να παραμβαίνουμε γέρος. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσα. Ελπίζουμε ότι θα βοηθούσα. Εμείς ε, είπαμε ότι ε, και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπλακεί όλα αυτά τα χρόνια. Ε, να σας πω ότι εσείς είχατε δύο μεγάλους πολέμους, αλλά δεν είχατε τόσους μικρούς πολέμους όπως συμβαίνουν εκεί. Εμείς θεωρούμε ότι ελπίζουμε ότι θα επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Όμως, ναι, φυσικά, είναι σωστό αυτό που είπατε ότι καλύτερο είναι να σταματήσουν αυτές οι σειράξεις πριν να ξεσπάσουν και να αναπτύξουμε τέτοιες ικανότητες. Όμως θέλω να σας πω ότι η Ήπειρος καταβάλει προσπάθειες Όσο ο Πρόεδρος θα απαντήσει στις ερωτήσεις της κυρίας Γκόμας. Όμως, οι κανόνες, οι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με την ε, εκλογική διαδικασία υπάρχουν για την καταμετρήση των ψήφων, Υπάρχουν κανόνες που λένε ότι η καταμέτρηση των ψήφων πρέπει να γίνει στα εκλογικά κέντρα υπό την παρουσία των παρατηρητών, των αρμοδίων φορέων κτλ. Και στα αστυνομικά τμήματα αναρτώνται τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ε, όλοι αυτοί οι κανόνες, όμως η πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν. Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα ότι ζητήσαμε από την Αφρικανική Ένωση να συστήσει μια ομάδα παρακολούθησης και αναφερόμαστε περισσότερο στον όρο monitors παρά observers. Γιατί είχαμε αυτό τον κωδικά διοντολογίας που συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ομάδα ανθρώπων που θα παρευρεθούν εκεί για να συμβάλλουν στο ότι θα τηρηθεί και ο νόμος αλλά και αυτός ο κώδικας διοντολογίας. Αν κάνω λοιπόν εγώ κάτι λάθος, αν δεν σεβαστώ δηλαδή τον κώδικα και την νομοθεσία, κάποιος μπορεί να πάει σε αυτή την ομάδα παρακολούθηση και να πει «Α, αυτός ο άνθρωπος έχει δράση λανθασμένα. Έτσι λοιπόν ε, θα μπορούσε να παρέμβει εκείνη τη στιγμή η ομάδα παρακολούθησης ε, προκειμένου να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που θα μπορέσουν να παρέμβουν και να δημιουργήσουν αυτό το καλό κλίμα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Euh, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησα, να προσθέσω και εγώ σε αυτά που είπατε. Γιατί οι, οι Αφρικανοί δεν καταφέρνουν να σταματήσουν τις τραγωδίες εγκαίρως. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρος Εμπέκη, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και ένα στοιχείο που επιτρέπει να καταλάβει κανείς το γιατί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε τη δυνατότητα διαχείρισης των κρίσεων και των συγκρούσεων σε μια προοπτική ιστορική και την έκρηξη αυτών των συγκρούσεων. Η Αφρική είναι μια ήπειρος, νέα ήπειρος. Όσον αφορά την οικοδόμηση εθνών, εννοώ, κρατών. Αυτό που συμβαίνει Δες, αυτά που συμβαίνουν δεν δείχνουν ότι είναι πιο βίαιοι πληθυσμοί του κόσμου οι Αφρικανοί. Αλλά πώς εξηγείται, είμαστε νέες χώρες, πολλές από τις χώρες αυτές δεν έχουν πετύχει την απαραίτητη σταθερότητα, προσπαθούν να πετύχουν σταθερότητα και αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται και χρόνο σε άλλες υπήρους. Δεύτερον, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, η δυνατότητα διαχείρισης των συγκρούσεων και αυτό χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτή η δυνατότητα και ξεκινήσαμε μέσω της Αφρικανικής Ενώσεως και άλλων περιφερειακών οργανισμών να αναπτύξουμε αυτή τη δυνατότητα διαχείρισης των κρίσεων. Αυτή η τραγωδία που δυστυχώς σήμερα λαμβάνει η χώρα υπάρχει, αλλά και οι Αφρικανοί είναι αυτοί που συμβάλλουν να σταματήσουν αυτά, παρόλο που είναι πολύ αργά, το γνωρίζουμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό το δυναμικό, αυτή τη δυνατότητα και είμαι σίγουρος ότι τελικά οι Αφρικανοί θα έχουμε, όπως και οι άλλοι, τη δυνατότητα, επαρκή δυνατότητα να διαχειριζόμαστε την ειρήνη και την ασφάλεια στην ε, Ήπειρό μας. Τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα των εκλογών στο Σουδάν, θα ήθελα καταρχάς να υπενθυμίσω το πολιτικό πλαίσιο. Από την ανάλυση μας όσον αφορά τον Νταρφούρ, ε, διαπιστώσαμε ότι η μακροπρόθεσμη λύση των προβλημάτων του Σουδάν πρέπει να εξευρεθεί στην ε, δημοκρατική μεταμόρφωση αυτής της χώρας. Αλλά αυτή η μεταμόρφωση δημοκρατική της χώρας χρειάζεται χρόνο. Ε, δεύτερο στοιχείο, οι εκλογές που προετοιμάζονται σήμερα αποτελούν κομμάτι της συμφωνίας, της Γενικής Συμφωνίας μεταξύ Βορρά και Νότου. Είναι ένα στοιχείο της συμφωνίας. Αυτές οι εκλογές λοιπόν θα πρέπει να λάβουν χώρα, να διεξαχθούν ε, στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Υπήρξαν πολλοί που ήθελαν να αναβληθούν οι εκλογές. Οι λαοί του Νότου, παραδείγματος χάρη, λένε όχι. Εμείς δεν δεχόμαστε αναβολή των εκλογών, διότι μια αναβολή των εκλογών σημαίνει αναβολή του δημοψηφίσματος, που είναι ο τελικός στόχος της Γενικής Συμφωνίας. Αυτές οι εκλογές λοιπόν θα πρέπει να λάβουν χώρα. Εν συνεχεία θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η χώρα εδώ και 25 χρόνια δεν έχει γνωρίσει εκλογές. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν, οργανωτικά προβλήματα. Η Εθνική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εκλογών υπάρχει, προβλέπεται από τον νόμο αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε η δουλειά της να είναι τέλεια. Υπάρχουν κενά, τα πολιτικά κόμματα μας ανέφεραν σαφώς την ύπαρξη κενών. Ο ρόλος μας, όπως είπε και ο πρόεδρος Εμπέκη, είναι να βοηθήσουμε ούτω ώστε οι εκλογές στο Σουδάν να διεξαχθούν ελεύθερα, δημοκρατικά και να συμμετάσχουν στο βαθμό του δυνατού οι περισσότεροι εκλογείς και να συμβάλλουμε όσο γίνεται από την πλευρά μας να επιληθούν τα προβλήματα με εξεκλογικής επιτροπής και των ε, πολιτικών κομμάτων. Ε, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα. Τώρα όσον αφορά τους παρατηρητές, προβλέπεται πράγματι να υπάρχουν εθνικοί παρατηρητές και η κοινωνία των πολιτών στον Νότο βοήθησε πολύ να υπάρξει κινητοποίηση όσον αφορά επιτήρηση των εκλογών. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει εξωτερικέ, όπω το κέντρο Κάρτερ και άλλοι φορεί, συνέβαλαν στην ε, προετοιμασία ε, της κοινωνίας των πολιτών. Στο βορρά το ίδιο. Θα υπάρξουν παρατηρητές εθνικοί και διεθνείς ε, παρατηρητές. Η Αφρικανική Ένωση, όπως ανέφερε ο Προέδρος, αποφάσισε να αποστείλει πρώτα απ' όλα τους monitor όπως αποκαλούμε, τους επόπτες που είναι ενδιάμεση αν θέλετε μεταξύ πολιτι... μεσάζοντες μεταξύ της Επιτροπής και πολιτικών κομμάτων, μεταξύ κυβερνήσεως και πολιτικών κομμάτων και μια σημαντική ομάδα παρατηρητών και άλλες αφρικανικές χώρες όπως η Νότια Αφρική όπως ε, οι χώρες μέλη του ΙΓΚΑΤ αποφάσισαν να αποστείλουν πολλούς παρατηρητές θα γίνει η επιτήρηση, θα υπάρχουν παρατηρητές και πιστεύουμε ότι αυτή η επιτήρηση θα αφορά όλη την διεξαγωγή των εκλογών. Είναι εδώ και μήνες πολλοί από τους παρατηρητές, διότι σήμερα γνωρίζετε ότι έχουν την, έχουμε την προετοιμασία, την προεκλογική περίοδο, προετοιμασία, ψηφοφορία, ημέρα εκλογών, καταμέτρηση ψήφων, αλλά και η περίοδος ακολουθεί πρέπει να επιτηρείται. Παρά αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Μπασίρ, θα υπάρχουν παρατηρητές, είναι ήδη εκεί οι παρατηρητές και θα κάνουν τη δουλειά τους. Επισκεφθήκαμε επανειλημμένα την Εθνική Επιτροπή των Εκλογών και μας εγγυήθηκε επανειλημμένα η Επιτροπή αυτή ότι οι παρατηρητές θα κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω λοιπόν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Σουδάν. Ίσως να μην είναι τέλειες, νομίζω ότι θα είναι όμως σημαντικό βήμα στο δρόμο του εκδημοκρατισμού της ε, χώρας αυτής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όπως βλέπετε και οι ίδιοι μόνοι σας, έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας και έχουμε κατάλογο έξι μελών που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Παρακαλώ να ε, επικεντρωθείτε και να υποβάλλετε το ερώτημά σας σε ένα λεπτό και θα παρακαλέσουμε τον πρόεδρο Μπέκη να απαντήσει και να ολοκληρώσει αυτή την συνεδρίασή μας. Πιστεύω είναι πολύ ενημερωτική και γι' αυτό μπαίνουμε στον πειρασμό να υποβάλλουμε περισσότερες ερωτήσεις και να ανακαλύπτουν περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Γκάλερ για ένα λεπτό πρώτος. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Εγώ Πώς αξιολογείτε ότι οι εμπλεκόμενοι, πόσο θεωρείτε ότι είναι δεσμευμένοι στη διαδικασία και στο εξωτερικό και στο εξωτερικό όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών γιατί ίσως και οι δύο πλευρές ε, θα θεωρήσουν πως έχουν ενισχυθεί ο καθένας ε, στο εκλογικό του κοινό δηλαδή ο πρόεδρος του Νότου θα πει ναι έχω εντολή για να περάσω στο δεύτερο γύρο ίσως για να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να διαχωριστούμε και μετά υπάρχει η Διεθνή κοινότητα και η Αφρικανική Ένωση. Δηλαδή η Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να καταλήξει στο εξή ότι θα αλλάξουν για πρώτη φορά τα σύνορα από την ανεξαρτησία. Θεωρείτε πως ε, θα παίξει ρόλο στο δεύτερο μέρος ε, η Αφρικανική Ένωση. Και ο Αραβικός Σύνδεσμος ε, τι ρόλο θεωρείτε ότι μπορεί να παίξει πολιτικά και οικονομικά για να παραμείνει και το Σουδάν και ο Πρόεδρος ε, στο πλαίσιο αυτό των εξελίξεων. Σας ευχαριστώ και εσείς για ένα λεπτό. Κύριε Μπέκη, θα αναφερθώ και εγώ σε αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφο κύριος Γκάλερ για το τι θα γίνει μετά τι εκλογέ. Ε, το δημοψήφισμα που θα γίνει του χρόνου. Τι ακούτε από τις δύο πλευρές ε, και από την κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Εάν έχουμε ανεξαρτησία η κυβέρνηση Μπασίρ ή η νέα κυβέρνηση θα την αποδεχτεί και στο Νότο Εάν δεν υπάρξει ανεξαρτησία, τι, τι θα γίνει. Κατόπιν, για τον Νότιο Σουδάν επίσης, η χώρα έχει πετρέλαιο. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους της σύγκρουσης. Ο ρόλος των πετρελαϊκών εταιριών γνωρίζω πως είναι οι Μαλαισιανές, Κινέζικες και εγώ πριν από 8 χρόνια είχα εμπλακεί με μία αυστριακο-σουηδική εταιρεία. είναι εταιρείε αυτέ, αλλά έχουν πολιτική επιρροή. Τι ρόλο παίζουν. Ευχαριστώ, η κυρία Σαμπίνε Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Μιλήσατε, κύριε Μπέκη, στην αρχή για τον ρόλο της κατανομής του πετρελαίου. και πάντα εκεί καταλήγει η λύση στα έσοδα του πετρελαίου. Πολλοί σχολιαστές λένε πως θα μπορούσε να βρεθεί και μία λύση μετά τον ε, διχασμό. Το βρίσκεται ρεαλιστικό. Μήπως η λύση είναι προϋπόθεση για να δεχτεί η κυβέρνηση την αποχώρηση του Νότου. Δεύτερον, πώς ε, βλέπετε το θέμα αυτό σε σχέση με τον νότο της Ιεμένης. Εάν αποσκυρτήσει ο νότος, μήπως αυτό θα δημιουργήσει, ο νότος Ιεμένης θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και για τον Ταρφούρ. Και κάτι ακόμα για τον Ταρφούρ. Στην ε, έκθεση της Αφρικανικής Ένωσης ζητάτε περισσότερα στρατεύματα του ΟΗΕ Στο Κονγκό, ας πούμε, υπάρχουν 20.000 στρατεύματα του ΟΗΕ και δεν επαρκούν. Αναφέρατε το ζήτημα φτώχεια πλούτος που πρέπει να λυθεί και νομίζω έχετε γράψει και στην έκθεσή σας το πρόβλημα του αναδασμού και της γης. Αυτό δεν λύνεται με στρατεύματα. Ευχαριστώ, κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι Σλοβένος γιατί... Ε, σωστό λέω γιατί μάλλον δεν έχετε ξανακούσει ποτέ τη Σλοβενική. Κύριε Μπέκη, έχετε την εντύπωση πως ε, όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής ε, για την προετοιμασία των εκλογών έχουν συμπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους και τους ενόπλους. Εγώ ήμουν στην Αμπούτζα παρατηρητή των εκλογών. Οι άνθρωποι, οι ένοπλοι, έχουν μεγάλη σημασία. Αυτοί πρέπει να δεχτούν να λάβουν δημοκρατικέ αποφάσει και η απόφασή του είναι εξίσου σημαντική με την απόφαση του κυρίου Μπασίρ για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών. Ένα άλλο ερώτημα. Τι γίνεται με τα ξένα συμφέροντα στο Σουδάν, ειδικά στον Ταρφούρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κριστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις πολύ σύντομες. για τις εκλογές. Νομίζετε ότι υπάρχει και πιθανότητα να μην υλοποιηθούν οι εκλογές και τελικά να γίνουν οι εκλογές ποιος θα υποφεληθεί. Ο πρόεδρος Μπασίτη τελευταία έχει αλλάξει στάση, από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει ύφος. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιος θα υποφεληθεί από εκλογές που θα γίνουν πολύ νωρίς αν υπάρχουν ε, εντάσεις. Η κυρία Λισαγερ Κοντσάρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ προκειμένου να αποτρέψουμε μελλοντικέ κρίσεις στην Αφρική, στο Σουδάν και σε άλλες ε, χώρες της Αφρικής. Θα ήθελα να ρωτήσω πώ ε, αξιολογείται τα νέα ότι η Κίνα, πολλές ευρωπαϊκέ χώρες, ευρωπαϊκές ε, εταιρείε αλλά και πολλά επενδυτικά τα μία ε, έχουν από κοινού αγοράσει γη στην Αφρική. Φαίνεται ε, ότι πρόκειται για δεύτερη ε, απόπειρα κατάκτηση της Αφρικής κατά κάποιο τρόπο. Πώς σχολιάζεται αυτό. Ευχαριστώ. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Μπαϊκή να απαντήσει. Μικρόφωνο παρακαλούμε. I, I hope, I hope we've taken them down. Ελπίζω να σημείωσα σωστά τις ερωτήσεις σας. Ανέφερα νωρίτερα ότι εργαστήκαμε επί ενός εγγράφου ενός κώδικα δεντολογίας για τις εκλογές. Κάποια μέρη το έχουν υπογράψει, το NCP, το LSPM και άλλα μέρη. Αλλά προετοιμάσαμε και ένα άλλο έγγραφο για να ασχοληθούμε με την ερώτηση που θέσετε. Αυτό το εγγραφό ονομάζεται «Διακήρυξη επικοινών δεσμεύσεων». Έχει να κάνει με δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα διάφορα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν και για τις εκλογές αλλά και για τον Ταρφούρ και για τη CPA. Έτσι λοιπόν, ποιο και είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχει μια κοινή δέσμευση όλων των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει μια εθνική συνένεση ότι αυτό πρέπει να γίνει σε σχέση με την επίλυση της σύραξης στον Ταρφούρ, αυτό πρέπει να γίνει για το δημοψήφισμα, τη συνέβηση του δημοψηφίσματος κτλ. Ανεξαρτήτως των εκλογών. δεν μπορούμε να πούμε ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Επομένως, γι' αυτό συντάξαμε αυτό το έγγραφο. Υπάρχει λοιπόν κοινή δεσμευσή μεταξύ των πολιτικών ηγετών στο Σουδάν για αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν το Σουδάν. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι το λένε αυτό ρητορικά, θεωρητικά και δεν υπάρχει πραγματική δέσμευση, αλλά υπάρχει μια κοινή βάση όπως σας είπα και αντικατοπτρίζεται αυτό στο έγγραφο που σας ανέφερα. Και νομίζω ότι η διεθνή κοινότητα θα συμφωνήσει με αυτό. Συνεργασόμαστε πάρα πολύ στενά με την Λίγκα των Αραβικών Κρατών. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε στο Κάιρο με τη Λίγκα και μας είπαν ε, ότι η των Αραβικών Κρατών θα ακολουθήσει την ε, ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι το έχουμε προσεξεί παρκώς το θέμα αυτό. Καλή στη χώρα λένε, στο πλαίσιο αυτών των κοινών δεσμεύσεων, ότι είναι απαραίτητο να σεβαστεί να δούμε όλες τις ε, διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στη CPA, στην Καθολική Ερνευτική Συμφωνία και πρέπει να υλοποιηθεί και το δημοψήφισμα έτσι όπως έχουμε σχεδιάσει και να σεβαστούμε και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Ο πρόεδρος ε, Μπασίρ στην προεκλογική εκστρατεία επέμεινε επί της ανάγκης να σεβαστούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ακόμη και αν ο λαός του Νοτιού Σουδάν αποφασίσει υπέρ της ανεξαρτησίας. Νομίζω όμως ότι υπάρχει γενική συμφωνία επ' αυτού, γιατί δεν θεωρώ ότι κανείς ε, στο Σουδάν θέλει να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Γιατί αν ε, κάποιος ε, μπλόκαρε τη διαδικασία, αν έλεγε ότι θα σταματήσουμε ουσιαστικά την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν, αν ήταν αυτό το αποτέλεσμα του ψηφίματο, τότε θα προκαλούσε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογές και όλοι έχουν τοποθετηθεί ειλικρινώ. Δεν ξέρω για τον πολιτικό ρόλο των πετρελαϊκών εταιριών. Πραγματικά δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείε. Στο πλαίσιο του μηχανισμού της Καθολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας ε, προβλέπεται να αναφέρουν τα στοιχεία περί της παραγωγής τους, περί του επιμερισμού των εισόδων από το πετρέλαιο. Όμως για τον πολιτικό ρόλο δεν ξέρω. Τώρα για το θέμα του καταμερισμού των εσόδων από το πετρέλαιο. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα διευθυντηθούν μετά το δημοψήφισμα. Στην πράξη του δημοψήφισματος για το Νότιο Σουδάν λέγεται ότι προβλέπεται από την νομοθεσία ότι πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα κατόπιν του τους και ένα από αυτά τα θέματα είναι το θέμα των εσόδων από το πετρέλαιο. Ήδη λαμβάνει λαμβάνουν χώρο κάποιες εργασίες για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή η παροχή διαβούλευση ε, συμβουλών με συγχωρείτε, και στα δύο μέρη για το πώς θα επιλύσουν αυτό το θέμα του επιμερισμού των εσόδων από το πετρέλαιο. Θα πρέπει να συνεχίσουν ε, και τα δύο μέρη τη συνεργασία στο τομέα αυτό. Έχουμε ουσιαστικά την παραγωγή στο νότο, αλλά όλη η αγωγή είναι στο βορρά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα αυτό, ανάλογα και με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όμως ήδη υπάρχει μια διαδικασία παροχή συμβουλών. Και νομίζω ότι η δέσμευση στο ότι ε, θα συνεχίσουν να μοιράζονται τα έσοδα από το πετρέλαιο είναι κάτι αναπόφευκτο. Τώρα αυτό που είπε ο προσβευτής Καμπάρη, το αναπληρωτής ε, του ειδικού επισταλμένου για τον Τερφούρ, είπε ότι θα πρέπει ε, να γίνει καταμερισμός των διαφόρων αρμοδιοτήτων στον Τερφούρ. Ε, ό,τι αφορά τη δύναμη την ελευτική δύναμη του ΟΗΕ, δεν υπάρχει τώρα ειδικό αίτημα για αύξηση. Νομίζω ότι υπάρχουν 20.000 ε, ε, μια δύναμη 20.000 δυνάμεων ε, από το στρατό και στην αστυνομία και υπάρχουν και 5.000 πολίτες. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αποφασισμένος ότι θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους εκεί. για αυτή τη δυνατότητα που αναφέρατε ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόβλεψη τίποτα. Δεν μας δείχνει τώρα ότι θα ακυρωθούν οι εκλογές για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι θα υλοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες ε, των εκλογών, την προετοιμασία των εκλογών. ο εκλογικό νόμος ε, ρυθμίζει το θέμα της σύνθεσης των εκλογικών επιτροπών κτλ. Αυτά τα ζητήματα ρυθμίζονται μέσω του κοινοβουλευτικού συστήματος. Φυσικά, βέβαια, στο κοινοβούλιο δεν συμμετέχουν οι ένοπλε δυνάμεις. Αυτές οι ένοπλες με συγχωρείτε. Και τη στιγμή που προετοιμαζόταν το Σουδάν για τις εκλογές, μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, όπως σας είπα, δεν είμαι σίγουρος ότι οι ένοπλες ομάδες είχαν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία. Ήταν έξω από τη διαδικασία λοιπόν. Αλλά προφανώς δεν θα μπορούσαμε να πούμε ας αφήσουμε τη διαδικασία προετοιμασίας των εκλογών ε, σε κρεμότητα μέχρι να είναι έτοιμες ε, οι ένοπλες ομάδες να συμμετέχουν στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν ε, αποκλείστηκαν αυτές οι ομάδες γι' αυτό το λόγο. Όμως τα διάφορα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν θεωρούν ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός. Τέθηκε και μια ερώτηση για τα ξένα συμφέροντα στον Ταρφούρ. Τι κάναμε εμεί ω πάνελ, ω ομάδα υψηλού επίπεδου. Είπαμε ότι ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Σουδάν, η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ακολουθήσει συνολικά την ίδια κατεύθυνση. Κάτι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό είναι το εξή. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διάφορες πρωτοβουλίες ε, αποκλίνουσες. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε όλοι μαζί. Εμείς τι κάναμε ως πάνελ. Διασφαλίσαμε ε, ότι συζητούσαμε τακτικά με τις όμορες χώρες έτσι ώστε να αναλαμβάνουμε δράση όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Και το ίδιο κάναμε και με τους ειδικού απεσταλμένους ε, της Ρωσίας, της Κίνας, ε, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει ξένη παρέμβαση στον Ταφούρο που ε, θέτει εμπλοκή στην επίλυση του ζητήματος. Νομίζω ότι υπάρχει συντονισμό σε διεθνές επίπεδο. Και Κάτι ακόμα. Το πάνελ μας ε, δεν έχει συζητήσει το θέμα της αγοράς γης στην Αφρική. Να σας πω ότι και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Γιατί άκουσα αυτές τις ιστορίες ότι άνθρωποι με πολλά χρήματα έρχονται και αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις γης. Εγώ ξέρω από παρελθούσα εμπειρία ότι τελικά σε χώρες όπου έγινε αυτό εμπόδισε την ανάπτυξη ότι παραδείγματο χάρη μπορεί μια χώρα να είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα δρόμο μέσα από αυτή την έκταση για να υπάρχει πρόσβαση σε, με εκείνε τι αγροτικέ κοινότητε. Και τελικά έρχεται ο γεωκτήμονα και λέει όχι, δεν μπορείτε να περάσετε το δρόμο μέσα από τη δική μου έκταση. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Όμως το πάνελ δεν ε, τα έχει συζητήσει αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο για την απόσχεση. Νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι η Πύρος είπε ότι το θέμα της ενότητας είναι σημαντικό και αν δείτε πώς είναι διαρθρωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αφρικανική Ένωση, με συγχωρείτε, προσπαθεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις δομές μας, Ούτε και εγώ ξέρω, παρεμβαίνει ο κύριος Πάσχου. Αλλά κοιτάξτε, οι φιλοδοξίες είναι οι ίδιες. Θέλουμε την ολοκλήρωση, η Αφρικανική Ενότητα κτλ. Παρά τον αντίστροφο. Αλλά εδώ μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες ε, ιστορικές συνθήκες στο Σουδάν, ε, στα πλαίσια των οποίων προκύπτει το ζήτημα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να πούμε με ποιο τρόπο θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαχείριση. Δηλαδή, ακόμη και να ε, υπάρξει διαζύγιο, είναι φιλικό. Να μην ε, αποτελέσει παράγοντα αστάθειας ε, και σύγκρουσης. Αν αποφασίσει να αποσχιστεί το Νότιο Σουδάν, να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε τη συνεργασία και την ολοκλήρωση. Προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, νομίζω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, πρέπει να σας χειροκροτήσουμε. Σας ευχαριστώ. And, ε, we all wish the people, you know. Και ευχόμαστε στον λαό του Σουδάν την καλή τύχη που χρειάζονται βεβαίω και την στήριξή σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, να σας ενημερώσω πως καταφέραμε να βρούμε άλλα 15 λεπτά. Με 11.30 ώρα θα έρθει ο κύριος ο Κάμπα. Οπότε έχουμε 20 ολόκληρα λεπτά για δύο γνωμοδοτήσεις. Και θέλω να προσπαθήσετε έτσι να τα καταφέρουμε γιατί τι κάνουμε, μια ημερήσια διάταξη δύο ημερών, τους σε μία. Αν το καταφέρουμε αυτό, ε, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι χωρίς ε, περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση. Ζητάω από την κυρία Νικόλ Κιλ Νίλσεν να μας πει την συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ κοινότητας και Πακιστάν. Λοιπόν, θα συντομεύσω λίγο την παρουσίαση, αλλά θα ήθελα να πάτε και στο λόγο και να μου πείτε τι θέλετε, ποια είναι η υποψή σας για τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα είπα τη συμφωνία η οποία συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη συνθήκη τη Αβώνας, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζετε. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι όσον αφορά το Πακιστάν, θα πρέπει να διερωτηθούμε σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υποδοχής αυτών των ανθρώπων σε μια χώρα η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση επί του παρόντος ε, θα ήθελα να αναφερθείτε όχι μόνο στις εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διότι το Συμβούλιο λέει ότι η πόρα απέχει από την ασφάλεια κατά στη χώρας και η γερουσία του Πακιστάν σε επίσημο έγγραφο αναφέρεται σε κάποιες πρακτικές βασανιστήριων που ακολουθούνται. Πολύ γρήγορα λοιπόν τα θέματα που τίθενται όσον αφορά την ασφάλεια σε αυτή τη χώρα ε, είναι εξαφανίσεις πάρα πολλές ανθρώπων, προβλήματα επιθέσεων κατά μειονοτήτων, εγκλήματα τιμής, ε, βιασμοί γυναικών, ε, βιοπραγίες κατά ομοφιλοφίνων, ε, η ποινή του θανάτου και τα βασανιστήρια. Αν εξετάσετε την συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πακιστάν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν έχουμε πολλά εχέγγυα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ερωτήματα που θέτουμε, ποια είναι τα εχέγγυα που εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων που επιστρέφουν θα γίνονται σεβαστά. Το Πακιστάν δεν υπέγραψε σημαντικέ διεθνεί συμβάσει όπω είναι η Σύμβαση τη Γενέβης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τουλάχιστον να θέσει κάποια χέγγια, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αντίθετα τι προηγούμενε προηγούμενες ε, συμφωνίες η ρήτρα μη συνεπιών δεν μπορεί να συμπεριληφθεί διότι να φέρει ρήτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα στα διεθνή κείμενα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν έχει υπογράψει το Πακιστάν αυτέ τι συμβάσει, δεν βάλαμε αυτή τη ρήτρα οπότε και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα και τώρα εν γέννη η συμφωνία ε, θέτει όλη την ευθύνη επί των κρατών λέγοντας ότι τα κράτη είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν σωστές συνθήκες για την επανεισδοχή. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται μια συμφωνία ε, και που συνεπάγεται την ευθύνη της Ευρώπης όταν πρόκειται τελικά περί διμερών συμφωνιών επανεισδοχής που εφαρμόζονται. Γιατί η ευθύνη βαρύνει την Ευρώπη υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, ενώ δεν συμμετέχει ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στην εφαρμογή της συμφωνίας, ούτε την εποπτεία της εκτέλεσης συμφωνίας. 11 συμφωνίες επανεισδοχής ήδη έχουν υπογραφεί και εφαρμοστεί και μέχρι τώρα δεν έχουν δημιουργήσει κανένα, καμία μάλλον, δεν έχουν δημιουργήσει καμία αξιολόγηση. Ε, συνεχίζουμε προχωράμε χωρίς αξιολόγηση. Εδώ κλείνω και οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Το Κοινοβούλιο λοιπόν δεν μπορεί ούτε να τροποποιήσει ούτε να αλλάξει το κείμενο τη παρού συμφωνία. Θα πρέπει είτε να την επικυρώσει συμφωνία είτε να την απορρίψει. Θα ήθελα να σα ακούσω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι τι έχετε να μα πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σόγκουλ έχει το λόγο για ένα δίλεπτον. Δύο λεπτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μετά από εννέα χρόνια διαπραγματεύσεων ε, καταλήξαμε σε ένα όχι και πολύ φοβερό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε αν συμφωνεί και το Πακιστανικό Κοινοβούλιο με αυτή τη συμφωνία. Και η συνάδελφος μόλις είπε πως ε, αυτή βεβαιω είναι η ε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πως υπάρχουν περιπτώσεις στην Ένωση στη... στις οποίες πως ε, άνθρωποι κρατούνται στην φυλακή επιμέρες και δεν ξέρουμε τώρα με τη συμφωνία αυτή αν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ πέρα και έχουμε την εντύπωση πως γιατί υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις. Οπότε εντάξει με τις βελτιώσεις αυτές σας την κάνουμε δεκτή. Σας ευχαριστώ Μπρέτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν είναι σαφές ότι το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό και λεπτό θέμα. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη συζήτηση αυτή. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν είναι σημαντικό εταίρος της Ένωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και γενικά θα ήταν προτιμότερο να έχουμε ένα πολύ σαφές πλαίσιο συνεργασίας για την επανεισδοχή. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα πλαίσιο παρά να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη θα δέχονται την επανεισδοχή περίπτωση Σε ένα τέτοιο σενάριο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να έρθει λόγο. Έτσι λοιπόν δεν θα υπήρχε δυνατότητα να εκφράσει αμφιβολίες σε σχέση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ λεπτό το θέμα φυσικά, αλλά μετά από έτη διαπραγματεύσεων έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι τελικά έχει γίνει κάποια πρόοδος και τελικά και τελικά θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα στα πλαίσια της Συμφωνίας Επανεσδικής. Ευχαριστώ. Τάνοκ. Η ομάδα μας θα υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω εάν διαβάσατε στον τύπο την τραγική περίπτωση ενός Βρετανού, ενός αγοριού πακιστανική καταγωγής που απήχθη στο Πακιστάν από ένα δίκτυο που έφτανε από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία και δύο ύποπτοι πακιστανικής καταγωγής κάτοικοι Ισπανίας ζήτησαν διερμηνέα ενώπιον του δικαστηρίου. Εν πάση περιπτώσει τώρα έχουν συλληφθεί μαζί με την ε, Ρουμανίδα σύζυγό τους και κατηγορούνται στο Πακιστάν. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το θέμα, είναι διεθνής. Η εγκληματικότητα χρειάζεται ε, η συμφωνία αυτή για τους διεθνείς εγκληματίες και για τους ε, υποαπέλασιν ε, εγκληματίες που απελευθερώνονται από την φυλακή. Βεβαίως το Πακιστάν δεν έχει και τα φοβερότερη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ ασκώ ειδικά κριτική όσον αφορά τις σχετικές μειονότητες όπως οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί, οι Ινδουιστές και τα δικαιώματα των γυναικών δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Επιτρέπεται επίσης και σε τζιχαντιστές να εκπαιδεύονται και ξεκινάνε και επιθέσεις προς την Ινδία από την επικράτεια του Πακιστάν. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα βεβαίως δεν αποτελούν λόγο να μην υπογράψουμε τη συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν. Οπότε η ομάδα μας ε, θα υποστηρίξει την συμφωνία αυτή επανεισδοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λόιζινγκ. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μια γενική κριτική σε αυτή την ε, συμφωνία. Εδώ πέρα πάλι το θέμα είναι πρώτα απ' όλα κατά βάση για ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από το Αφγανιστάν. Πολεμάει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, ή συμμετέχουν οι χώρες της και άλλες ε, χώρες, ε, άλλοι άνθρωποι εκδιώκονται. Και, να λύσουμε, και προσπαθούμε μετά να λύσουμε αυτό το, το πρόβλημα. Και υπάρχει βεβαίως και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι κάνει η Κομισιόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών που θα επιστρέψουν στο Πακιστάν. Τι προσπάθειες έχει αναλάβει. Ειδικά όσον αφορά και ανθρώπους οι οποίοι διαφεύγουν από το Αφγανιστάν. Είναι γνωστή η κατάσταση στο Πακιστάν, ειδικά η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ε, οργανώσεις ε, ασκούν κριτική. Να αναφερθώ τώρα στο πρόβλημα της συλλογικής ε, απέλασης. Γιατί οι άνθρωποι μαζεύονται σε κάτι άθλια κέντρα υπό άθλιες συνθήκες και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και ένα ερώτημα ακόμα. Γιατί στη μεικτή αυτή η επιτροπή δεν υπάρχουν ε, μήκυο για να επιτηρήσουν την, ε, ε, συμφωνία. Αυτή είναι μια κατάσταση που ενοχλεί τις μη κυβερνητικέ αυτές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο κύριος Μπουσακεβίτς από την Κομισιόν. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις απόψεις που ακούστηκαν. Καταρχήν αναφερθώ με συντομία Ωστόσο, υπόθηκαν για τι ελλείψει τη διασυμφωνία συμφωνία ό,τι αφορά τον non-affection αυτή τη σχετική ρήτρα. Ε, υπάρχει η ρήτρα αυτή, δεν είναι τόσο εκτεταμένη ω συνήθω, αλλά υπάρχει στο άρθρο 15. Εκεί γίνεται αναφορά ότι είναι υπό ότι είναι επιφύλαξη η συμφωνία αυτή βάσει των ευθυνών του Πακιστάν προκίνων από το διεθνέ δίκαιο. Τώρα, το, αν αναλαμβάνουμε τι αντίστοιχε ευθύνε μα ε, από νομική σκοπιά μιλώντα, δεν αλλάζουν και πολλά γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, υπογράψει ε, τη Συμβέση της Γενέβης και σέβονται και πρέπει να σέβονται τη Συνθήκη της Γενέβης. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έλεγχο, το δικό μας, τη συμφωνία φυσικά η Κοινή Επιτροπή Επενδυσδοχής ε, συμπεριλαμβάνει τη συμφωνία. Εμείς εκπροσωπούμε την Ένωση στην Επιτροπή αυτή. Μας ε, βοηθούν και τα κράτη-μέλη, μας επικουρούν τα κράτη-μέλη το αν υπάρχουν μη καπαόμικρον ή όχι. Θα μπορούσε κάποιο να το αναφέρει αυτό σε επιχείρημα, αλλά να σα επισημάνω ότι πρόκειται για μια διοικητική συμφωνία, δηλαδή αφορά τη συνεργασία μεταξύ διοικήσεων. Και τώρα έρχομαι και στο κύριο θέμα. Πώς σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία δεν ε, αφαιρεί τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη υπό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό το διεθνές δίκαιο. Έχουμε τις ε, οδηγίες ε, περί της υποδοχής, έχουμε συμφωνίες, οδηγίες, με συγχωρείτε, για την προστασία των προσφύγων. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να υποστηρίξετε τη συμφωνία. Φυσικά καμία νομική πράξη δεν είναι τέλεια, αλλά εδώ συζητούμε περισσότερο για την ορθή εφαρμογή όλου του συστήματος, δηλαδή και το σύστημα του ασύλου, της διεθνούς προστασίας κτλ. Αυτό είναι το πραγματικό νομικό περιεχόμενο της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ξέρετε ότι η κυρία Κιλ Νίλσεν έλαβε την ε, απάντηση, αλλά θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε, να συνοψίσετε. Ακούστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω την απάντηση απολύτως, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ε, έχουμε εδώ ανάληψη ευθύνη ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν υπάρχουν εγγυήσει στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να δοθούν οι εγγυήσει αυτέ. Αν υπάρξει αυτή η συμφωνία, θα πρέπει να απαντήσουμε στα θέματα που τέθηκαν Δηλαδή αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτή την παρακολούθηση που δεν ε, κάνουμε σήμερα. Δεν υπάρχει αυτή η παρακολούθηση, αυτή η συνέχιση και δεν υπάρχουν εγγυήσει. Σαν ε, εμπλακή Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε και αυτό το θέμα. Εγώ αυτό το κύριο θέμα θέτω δηλαδή την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις σχετικές εγγυήσεις. Αναφέρθηκα και το θέμα των Αφγανών, ξέρετε ότι η πρώτη φράση λέει η σύναψη συμφωνίας επανεισδοχή με το Πακιστάν ανήκει στα μέτρα που συστήνονται στο πλαίσιο δράσης του Αφγανιστάν που παρουσιάστηκε το 99. Έτσι λοιπόν, ε, εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένες επιστροφές ε, από Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, Αφγανών και υπήρξε πρόβλημα γιατί τα έγγραφα για την επιστροφή δεν ήταν ικανοποιητικά, ε, δεν υπήρχαν εγγυήσεις από τον νόμο για τα δικαιώματα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Αφγανών. Ναι, ξέρω ότι μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση και με τους άλλους και οδούς και με την Κομισιόν για να διευκρινίσετε αυτά τα προβλήματα που εκκρεμούν. Και τώρα, να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω, θα ζητούσα από τον κύριο Μπιέλλαν να μας παρουσιάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και το ρόλο των μακροπεφεριών στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση για το ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής ε, έχει εκπονηθεί και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία το 2006 και τώρα συνεισφέρει στην εφαρμογή της. Η Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που είναι αρμόδια για την εφαρμογή το εξετάζει το θέμα από τη σκοπιά της ανάπτυξης της περιοχής της Βαλτικής θάλασσας ο δικός μας ε, ο ρόλος ε, είναι να προσδώσουμε μια διεθνή διάσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι εδώ ο πιο σημαντικός εταίρος είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Χωρίς ε, συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία η εφαρμογή της στρατηγικής δεν θα είναι δυνατή μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχω τονίσει αυτό στην γνωμοδότησή μου σε πάρα πολλά σημεία και επίσης ε, έχουν ενεργοποιηθεί 220 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. οι πόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, μόνο για εξωτερικές δράσεις στην περίπτωση αυτή. Θέλω να ενθαρρύνω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για να δούμε μήπως ε, θα πρέπει αυτά τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα χρησιμοποιήσουμε και στα πλαίσια του 2011. Επίσης, έχουμε κάποιες προκλήσεις ε, που πρέπει να σκεφτούμε, όπως ε, το θέμα της ενέργειας, το project North Stream. Σε συνεργασία με τη Ρωσία πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας ε, όταν θα συνάψουμε νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία. Δεν ε, μπορούμε να ξεχνούμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν ε, συζητούμε το θέμα της συνεργασίας με τη Ρωσία στο θέμα της Βαλτικής θάλασσας. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε. Περιμένω τα δικά σας σχόλια και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες, για την κατάθεση τροπολογιών ε, είναι στις 25 Μαρτίου 12 το μεσημέρι, αυτό επειδή ε, έχουμε ε, πολύ εντατικό πρόγραμμα τον Απρίλιο και ε, λόγω του φόρτου εργασιών θα σας παρακαλούσα στα αγγλικά να μας καταθέσετε τις τροπολογίες. Μάλιστα, 25 Μαρτίου είναι η προθεσμία στις 12 το μεσημέρι. Τώρα... Έχουμε περίπου πέντε αγορητές που το λόγο. Κύριος Κάμπο θα πρέπει να έρθει εδώ Κατέφτασε ήδη ο κ. Σοκάμπο. Λοιπόν, πραγματικά, πραγματικά σας το λέω, να τηρήσετε τα όρια. 30 δευτερόλεπτα. Ή κάτι παρεμφερές. Κύριε Μίρσκι, έχετε το λόγο πρώτος. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, θα ήθελα να θέσω κάτι εκ μέρους της ομάδας μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο εισηγητής ακολούθησε πολύ επικοδομητική προσέγγιση, ακολουθεί σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θέλω να περιοριστούμε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία ωφέλησαν όλους τους κατοίκους της περιοχής της Βαλτικής και θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε οι εσδήποτε δραστηριότητες που θα επέτρεπαν να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Ρωσία επί αμοιβαίας εποφελούς βάσεως, αμοιβαίως εποφελούς βάσεως. Ξέρετε ότι ε, κατασκευάζεται ο γογός φυσικού αερίου ε, Nord Stream. Γιατί δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πρόγραμμα. Μόνο η Γερμανία θα πάρει ενέργεια από αυτό τον αγωγό. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα κράτη της Βαλτικής. Ε, Πώ ταιριάζουν στην εξίσωση. Αυτό οφείλεται ότι δεν συμμετέχει η Ευρώπη συνολό τη σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον συγκεκριτή για το κείμενο, το υποστηρίξουμε. Πάρα πολύ σύντομα, λέει ο Πρόεδρος. επόμενο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Υπάρχει ένα προβληματάκι για την Επιτροπή μα. Είναι ότι η στρατηγική για τη Βαλτική θεωρείται εσωτερική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Κατά ανάγκη θα εμπεριέχει και εξωτερικές πτυχές λέει ο κ. Αναγνωρίζω όμως τον άριστο ρόλο του συναδέλφου Μπίλαν. Το άρθρο 1 με προβληματίζει. Μπορούμε να το πούμε, να το διατυπώσουμε ούτως ώστε να λέω ότι η εσωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει επικοδομητική συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Ε, το θέμα της βόρειας διάστασης επίσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτόν με σύγχρονους όρους. Οι εξωτερικές πτυχές όμως της στρατηγικής αυτής θα συμπεριλαμβάνουν αυτό που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εξασφαλίζεται η ασφάλεια ε, στην ε, περιοχή, και θα καλύπτονται και περιβαλλοντικές πτυχές και τα ποτάμια. Και η Λευκορωσία εισέρχεται στην εξίσωση. Μία εξωτερική πτυχή είναι η διακυβερνητική συνεργασία για την εφαρμογή και την υλοποίηση της στρατηγικής. Πρέπει να ειδωθεί ως θέμα συνεργασίας, να υπάρξει συνέργεια, να ενωθούν πόροι για υπερεθνικά προγράμματα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να σκέφτεται να προσεγγίσει το θέμα από την έποψη της βόρειας διάστασης. Ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο είχε δώσει ένα ειδικό κονδύλι 20 εκατομμύρια για φέτος ο συνάδελφος Μίνσκης είπε ότι για τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να επαναξετάσουμε το θέμα της χρήσης αυτών των χρημάτων για εσωτερική στρατηγική. Τέλος κύριε Πρόεδρε, η συμμετοχή της Ρωσίας και των άλλων εταίρων. Πρέπει να επιμείνουμε επίσης επικοινών ευθυνών και υποχρεώσεων. Παραδείγματο χάρη θα ήταν λογικό να αναφέρουμε εδώ ότι η Ρωσία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να, ε, να, να προσχωρήσει στη συμφωνία ΕΣΠΟ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. ο κ. Παλέτσκη, συντομότατα. Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις ε, προτάσεις του κυρίου Άνταμ και προτείνω δύο ακόμα παρατηρήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα για τη συνεργασία με το Καλίνιγκραντ την ε, περιοχή αυτή της Ρωσίας. Καλό θα είναι να το διατυπώσουμε έτσι ώστε να αποτελέσει η συνεργασία αυτή πιλωτικό έργο της Ένωσης για τη συνεργασία με τη Ρωσία. Ένα καλό παράδειγμα και τέλος θεωρώ πως πρέπει να αναφέρουμε την ανάγκη διευκόλυνσης του καθεστώτος θεωρήσεων με Ρωσία και Λευκορωσία. Σας ευχαριστώ εγώ κύριε Μπαλέτσκης, ο κύριος Λαντσμπέργκης. κοιτώντας ε, τις προτάσεις της Επιτροπής, προφανώς δεν ανησυχεί για τη Στρατηγική Επιτροπή, αλλά μόνο για το ρόλο της Ρωσίας και την πρόσβασή της στον ε, προϋπολογισμό της Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, απομακρυνόμαστε από το βασικό ζήτημα και πάμε στη βόρεια διάσταση. Στις δε προτάσεις, μία λέξη επαναλαμβάνεται συνεχώς. Το μόνο. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να αλλάξει αυτό που λέει στην πρώτη παράγραφο. Που λέει ότι τα σχέδια αυτά θα επιτύχουν μόνο. Όχι. Θα είναι πιο επιτυχή εάν έχουμε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Όχι μόνο εάν. Μετά λέει να υπάρξει μια επιπρόσθετη βάση αλλά η στρατηγική μας πρέπει να έχει μία βάση και όχι δεν είναι κάποια αυταξία το ίδιο και στην τέταρτη παράγραφο η στρατηγική της Βαλτικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εξωτερική δράση. Συνέχεια μόνο και μόνο, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα χωρίς τη Ρωσία. Εδώ έχουμε μονομέρεια. Εγώ θα προτείνω τροπολογίες που να λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγική και για εξωτερική δράση, όχι μόνο και μόνο. Δηλαδή έτσι που υπάρχει εδώ μέσα σημαίνει πως η χρήση των, των κονδυλίων της Ένωσης θα ε, ελέγχεται από τη Ρωσία. Ε, παραπάει. Με συγχωρείτε. Για την ώρα σας συγχωρούμε. Λοιπόν, η κυρία Γιάννερμάκη. Τρία σύντομα πράγματα. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με αυτό το οποίο έχει υποθεί και επαναλαμβάνεται και εδώ πέρα. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί 20 εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί μόνο για συνεργασία με τη Ρωσία. Αλλά αυτό είναι στην έκθεση της ε, Κομισιόν. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε ίσω να το κάνουμε έτσι κάπως πιο, πιο έντονο, για να χρησιμοποιηθούν και αλλιώ τα λεφτά. Κατόπιν. Κάτι άλλο που αφορά την πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένα βήματα και προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Μετά, όσον αφορά το σημείο 1. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούμε με τους εξωτερικούς εταίρους. Είναι κάτι άλλο από τις χώρες. Ε, να το πούμε πιο σαφώς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν επειδή έχουμε ήδη καθυστερήσει και έχουμε και έναν καλεσμένο. Θα ήθελα ο κύριος Μπιέλαν να έρθει σε επαφή μαζί σας και να τα συζητήσει αυτά τα ζητήματα και είμαι σίγουρος πως θα βρείτε μια λύση. Η προθεσμία, όπως είπα, είναι του Ευαγγελισμού στις 12 η ώρα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. Το οποίο είναι η Επιτροπή ε, συνάντηση με την και από την Υπό Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ καλωσορίζουμε τους κυρίους Δέβα και Χάουταλα. Και θέλουμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Λουίς Μαρενό Κάμπο, που είναι εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο πρώτος άνθρωπος που άσκησε αυτά τα καθήκοντα από την ίδρυση του δικαστηρίου το 2003 ο κύριος ε, Κάμπο έχει εμπειρία στην ε, εκδίκαση και άλλων ε, αξιόπινων πράξεων που διαπράκτησαν από τη δικτατορία στην Αργεντινή το 70 και το 80. Επίσης ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ και στο Πανεπιστήμιο του Μπένος Άιρες επικεφαλής ε, τώρα της ε, ΥΠΑ ε, θα ήθελα να πει δύο λόγια και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον κύριο ναι. Κάμπο και κατόπιν στον κύριο Τέβα. Ευχαριστώ. Είναι τιμή και χαρά μας που σας έχουμε εδώ κύριο Κάμπο, εκ μέρους της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν μπορώ παρά να τονίσω πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη στον τομέα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και πω τονίζουμε το θέμα του διεθνούς ποινικού δικαστήριου και το ρόλο του. Συναντήθηκα με τον αρχιδικαστή Σόγκ και θα έρθει στην υποεπιτροπή μα 24 Απριλίου ρω. και συναντήθηκα και με τον συνάδελφό σα στο δικαστήριο τον απειοτή δικαστή. Συζητήσαμε πρόσφατα την, το πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτές, το θέμα των μαζικών αυτών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φρικαλαιοτήτων σε μαζική κλίμακα. Πώς μπορεί να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προώθηση της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης ούτως ώστε να αποφύγουμε ε, τέτοιες ε, ομαδικές φρικαλαιότητες, ε, ε, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, έχουμε ε, την ε, ε, ανεξέταση της σύμβασης της Ρώμης και την έκθεση Κάμπαλα πάνω σε αυτό. Πώς πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει τα επόμενα βήματα, τα εξελεκτικά όσον αφορά το Διεθνές Δικαστήριο. Και τέλος, σας πω, θα σας πω πόσο σημαντικό θεωρώ ότι είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν οικονομικά το δικαστήριο διότι αξίζει περισσότερους πόρους από ό,τι διαθέτει. Με αυτά τα λόγια, καλώς ήρθατε εκ μέρους της Υποπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, καθώς όπως είπατε είμαι ο πρώτος αγγελέας που εργάζεται για σας. Εσείς ε, ουσιαστικά υιοθετείτε την νομοθεσία και εγώ πρέπει να διερευνώ ε, αυτές τις υποθέσεις και να σηκώ τις κατηγορίες. Όμως ο αντίκτυπος του δικαστηρίου εξαρτάται από εσά. Ουσιαστικά το δικαστήριο είναι το πρόσωπο, η όψη του συστήματος, αλλά η δύναμη του συστήματος ε, έγκυται στη δέσμευση δέσμευση των μερών και των διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να περάσω στο θέμα της πρόληψης. Σε αυτό που αναφερθήκατε, τα μαζικά εγκλήματα διαπράττονται για να δημιουργηθεί εξουσία και γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε ένα σύστημα πρόληψης των εγκλημάτων γιατί όταν ε, έχουμε τελικά δίωξη αυτών των ατόμων που διαπράττουν εγκλήματα τελικά δεν μπορούν να τα διαπράξουν πλέον και το καλύτερο παράδειγμα είναι η Κένια μετά τις εκλογές 2007-2008 στην Κένια υπήρξαν ε, μαζικές βιοπραγίες ε, Κοφιανάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στο να σταματήσουν αυτά τα εγκλήματα. Τώρα δεν θέλουμε να επανέλθουμε στη βία στι εκλογέ του 2012 και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασκηθεί έρευνα για αυτά τα εγκλήματα του παρελθόντος για την Κένια. Θέλουμε να αυξήσουμε την βεβαιότητα, την ασφάλεια. Γι' αυτό υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ισχυρή δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να, ξέρετε, ε, πρέπει να ξέρουν μάλιστα όσο διαπράττουν εγκλήματα ότι θα διωχθούν είτε εθνικά είτε σε διεθνέ επίπεδο. Και έτσι πρέπει να δράσουμε για να σταματήσουμε τα μαζικά εγκλήματα. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Αλλά εσεί ε, κατόπιν εγκρίνατε ε, αυτό το, η νομοθεσία στη Ρώμη πριν 11 χρόνια τώρα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε και νομίζω ότι αυτή είναι η κυρία ιδέα στην Καμπάλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι λειτουργεί το σύστημα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξή. Ε, στην Ευρώπη υπήρξαν βιοπραγίε πριν 60 χρόνια και μετά είχαμε και στα Βαλκάνια. Δεν υπήρξαν άλλε βιοπραγίε. Έτσι λοιπόν, ε, στην Ευρώπη μπορεί να έχει κλείσει το θέμα, αλλά στην Αφρική χρειάζονται υποστήριξη. Στην Κένια ήταν ενδιαφέρον το θέμα γιατί ο Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρο ε, μου είπαν δεν μπορούμε να ζητήσουμε τη δική σα παρέμβαση, αλλά θέλουμε να σα υποστηρίξουμε και βλέπουμε ότι πραγματικά και εκατοντάδε κράτη και το δικαστήριο συμβάλλουν στο να σταματήσουν βιοπραγίε στην Κένια. Έτσι λοιπόν, ε, το κύριο μήνυμα είναι, αλλά κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά πέρα από το ρόλο του δικαστηρίου χρειαζόμαστε και πολιτική ηγεσία. Αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντέβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μα ήταν συναρπαστική η παρέμβασή σας έτσι, σύντομη. Και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία μας είπατε. Κύρια Σίλβα το ανέφερε. Το εγώ το πάντα το, το ποινικό διεθνές δικαστήριο και τα ειδικά δικαστήρια τα θεωρούν πάντα μια διαδικασία συμφιλίωσης. Αλλά αυτό το οποίο μας είπε ο εισαγγελέα είναι πως το ποινικό δικαστήριο μπορεί να παίξει ρόλο αποτρεπτικό ορισμένων καταστάσεων. Μια νέα ιδέα την οποία καλωσορίζω προσωπικά. Γιατί επειδή είμαι και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, δίνουμε δισεκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων μας σε συγκρούσεις και καταστάσεις μετά τις συγκρούσεις και 5% αυτών των χωρών ξανακυλάνε στη σύγκρουση. Είναι φαύλος κύκλος. Εάν χρησιμοποιήσουμε όμως ως απειλή το Διεθνές Ποινικό ε, Δικαστήριο, ως ε, δαμόκλειο σπάθη, τότε παίζει πλέον ένα ρόλο αποτροπής που το Κοινοβούλιο νομίζω μπορεί να αγκαλιάσει, Όπως είπε και η κυρία Άρτολα. Μπορούμε να, να συνεργαστούμε σε αυτό. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει και ο Πρόεδρος. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε την Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Εισαγγελέα που ήρθατε. Να σας ρωτήσω, μόλις είχαμε μία συζήτηση για την οργάνωση των εκλογών στο Σουδάν και ο πρόεδρος ο κύριος Μπέκη που είναι επικεφαλής του πάνελ για το Σουδάν είπε πως ε, για τα θέματα δικαιοσύνης για τα εγκλήματα του Νταρφούρ, μία λύση είναι ένα υβριδικό δικαστήριο για να διώξει ε, νομίζω ζητήματα που δεν θα έρχονταν ενώπιον του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου. Οπότε έχουμε αφενός τις κατηγορίες που έχει απαγγείλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και από την άλλη έχουμε εγκλήματα που δεν θα πήγαιναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά θα απασχολούσαν ένα υβριδικό δικαστήριο με και εθνικούς δικαστές. Γνωρίζετε αυτή τη λύση θεωρείτε πως θα μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο το, το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο και θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Να σας ρωτήσω και κάτι, κάποια άλλα πράγματα. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομισιών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν ή και κρατών μελών στο να διασφαλίσουν πως ε, οι ύποπτοι, οι κατηγορούμενοι ναι, σύρονται ενώπιον του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Μπορείτε τέλος ε, να μας πείτε πού βρίσκεται η δίωξη για τα εγκλήματα πολέμου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Ευχαριστώ. I think it's very important. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα που παρουσιάσατε και το Κοινοβούλιο πρέπει να συζητήσει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αυτήν την εξωτερική εκπροσώπηση. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία, γιατί Όπω είπατε, η ιδέα να χρησιμοποιηθεί το δικαστήριο για προληπτικού λόγου ήταν μια ιδέα. Στην ε, Σύμβαση τη Ρώμη ε, είχαμε τέλο τη ατιμορρησία. Αυτό πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη Τη επιτέλεση νέων εγκλημάτων. Αυτό το θέμα της πρόληψης λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό νομίζω ότι και εσείς πρέπει να εμπλακείτε ε, στην ε, άσκηση τη εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι ο ρόλος του Πρέδου Μπέκη ήταν πολύ σημαντικό στον Τερφούρ και αυτό σε πίεση και αυτό τόνισε ότι χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη. Ε, όσο ο πρόεδρος Βασίλης στην εξουσία θα διαπράττει περαιτέρω εγκλήματα. Ε, μετά την επόμενη, την επόμενη μέρα της συμφωνίας επιτέθηκε, όπως ξέρετε, και εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες ε, πολίτες ε, στη Τζαρά Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό. Πρέπει να ακολουθεί μια συνεπή στάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο πρόεδρος Μπασίρ ε, και σήμερα και μετά τις εκλογές θα πρέπει να σεβαστεί τον νόμο και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ νομίζω ότι αν είστε συνεπείς τότε αυτό θα οδηγήσει και σε βεβαιότητα. Τώρα για την λαϊκή δημοκρατία του Κογκό, εδώ εργαζόμαστε πολύ καλά, ε, αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε ποια είναι τα κύρια εγκλήματα ε, που διαπράττονται εκεί, κυρίως ε, φιλετικού χαρακτήρα. Ενώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο όμως αυτό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Και ναι, το Βέλγιο συνέλαβε το Τσάμπουργκ σε μία μέρα και λέει το κοινοβούλιο είναι πιο περίπλοκη υπόθεση του Μπασίρ χάρη και γι' αυτό επανέρχομαι ε, στο θέμα των υπηρεσιών σας εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να χαράξετε μία πολιτική γιατί πρόκειται για μία νέα ιδέα, πρέπει να αναπτύξετε μία πολιτική για το πώς θα γίνεται διαχείριση αυτής της σύραξης σε επίπεδο διπλωματών. Ευχαριστώ. Κυρία Λόχπλη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Η σύνοδος ε, της ε, Καμπάλα βοήθησε στο να δούμε και τι λειτουργεί σωστά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο τι δεν λειτουργήσε τόσο καλά. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τη δική σας εκτίμηση. Τι θα μπορούσε να βελτιώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πού βλέπετε την δυνατότητα να σας στηρίξουμε. Κάτι το οποίο βλέπω και μου έκανε εντύπωση, υπάρχει δυνατότητα προγράμματος Προστασία μαρτύρων. Είναι σημαντικό να προστατευτούν τα άτομα, εάν καταθέτουν κατά των πρώην κυβερνήσεών τους. Και διάβασα πως σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μόνο στο γύρω 40% των προγραμμάτων αυτών ε, προσφέρουν ε, προστασία σε άλλες χώρες. Οπότε θα με ενδιαφέρε να μάθω πώς αξιολογείται ε, το τι μπορεί να βελτιωθεί στον τρόπο λειτουργίας του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ πολύ. Έχετε τον λόγο. Η έκθεση της Καμπάλα συμπεριλάμβανε τέσσερα σημεία, αλλά αφορούν το σύστημα όλο συνολικά, δηλαδή το πώς το σύστημα προστατεύει τα θύματα, τη συνεργασία με το δικαστήριο, αυτό το οποίο λέμε επίσης συμπληρωματικότητα, δηλαδή το πώς το δικαστήριο βοηθάει οι εθνικές αρχές και τέταρτον είναι η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα τέσσερα ζητήματα. Τα θύματα έχουμε, έχουμε καλή συνεργασία. Η συνεργασία πάει καλά επίσης. Η δύσκολος τομέας είναι οι συλλήψεις του Παγάντα, του Τζόζεφ Κόνη, του Πρόεδρου Μπασίρα. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Μετά υπάρχει το πρόβλημα της ε, συμπληρωματικότητας ε, ε, για να φερθώ και στις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης, γιατί η Ευρώπη κατά κανόνα προωθεί την εκπαίδευση δικαστών, αλλά στο Κονγκό υπάρχει Κογκολέζος δικαστής που καταδίκασε δύο άτομα που, καταδίκασε, που, βίασαν μία γυναίκα. Μετά πάνε στη φυλακή και στη δεν έχουν φαΐ. Οπότε οι φυλακέ μετά είναι ανοιχτέ, ανοίγουν τι πόρτε. Δηλαδή, τι να καταδικάζει κάποιον αν δεν μένει φυλακή. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο δικαστές ε, και εισαγγελίες, είναι ασφάλεια για τους ε, μάρτυρες και τους λοιπούς. Οπότε στις εξωτερικές σχέσεις πρέπει να αναπτύξετε το πώς θα υποστηρίξετε τις χώρες ε, στην όλη διαδικασία. Δεν είναι μόνο θέμα δικαστών, είναι θέμα ασφάλειας είναι να προστατεύσουμε τα θύματα. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, ναι, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να προστατεύσω τα, θύματα. Αυτό, αυτό κάνω κατά βάση. Είμαι υπερήφανος γιατί σε 7 χρόνια δουλειά. Ε, που ερευνήσαμε τέσσερα μαζικά εγκλήματα, κανένας μάρτυρας δεν, δεν επηρεάστηκε. Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Νομίζω μπορούμε να προστατεύσουμε δε τους ε, μάρτυρες ή στη χώρα τους ή σε γειτονικέ χώρες. Γιατί οι άνθρωποι στον Ταρφούρ θέλουν να μείνουν στον Ταρφούρ, δεν, δεν θέλουν να φύγουν. Οπότε δεν έχει νόημα να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα στην Ευρώπη. Τοπικά νομίζω είναι καλύτερα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Βεβαίω, εμένα η αρμοδιότητά μου στο δικαστήριο είναι άλλη, αλλά η προστασία των θυμάτων είναι σημαντική, αλλά στην Κένια, παραδείγματο χάρη σήμερα, η προστασία των, των απλών πολιτών δεν είναι ευθύνη δική μας, είναι της ε, κυβέρνησης Κένιας. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε την Κένια, το τι γίνεται σήμερα, το τι κάνει η αστυνομία για να προστατεύσει τον κόσμο. Γιατί ακούγεται πως η αστυνομία σκοτώνει τον κόσμο. Αυτό είναι παράδεκτο. Αυτό νομίζω μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε την κυβέρνηση το τι κάνουν με την αστυνομία, του στρατό κτλ. Και όπου βρουν λάθη να τα διορθώσουν. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια καταρχάς κύριε Σαγγελέφ για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η καριέρα σας. Εγώ είμαι από ένα εθνικό κόμμα, το, τους Βρετανούς συντηρητικούς που εξακολουθούμε να συμπαριστάμεθα στην αμερικανική θέση για τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ίσως ε, τελικά οι διώξεις του δικαστηρίου αυτού να έχουν πολιτικά κίνητρα. Μέχρι τώρα όμως το ιστορικό σας, κυρίως το δικό σας, σαν ε, επικεφαλής εισαγγελές, δείχνω ότι δεν ε, ακολουθείτε αυτή την προσέγγιση και χαιρόμαστε. Ένα, σε ένα κλίμα τιμωρησία συμφωνούμε όσον αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, γενοκτονίες είναι κάτι απαράδεκτο, κυρίως τώρα τον 21ο αιώνα όταν έχουμε αναπτύξει διεθνή νομολογία στον τομέα. Λοιπόν, το ερώτημα που έχω να σας απευθύνω είναι πώς θα πείσουμε τι μεγάλε δυνάμει τι Ηνωμένε Πολιτείε την Ινδία και την Κίνα με άλλα λόγια, επί παραδείγματι και άλλε χώρε όπω το Ισραήλ, τι πρώτε τρει που ανέφερα, Κίνα και ΗΠΑ, που παραδόξω συμφώνησαν τον κύριο Μπασίρ να τον παραπέμψουν στο Συμβούλιο ασφαλεία, παρόλο που δεν έχουν υπογράψει το σύμφωνο τη νόμη και δείχνει ότι είναι αμφιλεγόμενη η θέση του. Πώ μπορούμε να πείσουμε, λέω, την Αμερική και την Κίνα στην Καμπάλα να χαλαρώσουν και να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση τη Ρώμη όπω έχει τροποποιηθεί, ούτω ώστε να διασκεδαστούν ησυχίε. Απάντηση. Νομίζω ότι έχουν χαλαρώσει, αλλά δεν θα υπογράψουν τη συνθήκη αμέσω. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται, χρειάζεται χρόνο. Η Κίνα ε, δεν είναι ένα εταίρο που δεν υπογράψει. Η Ρωσία μας έστειλε 3.000 ανακοινώσεις ε, για τα εγκλήματα που διεπράξα στη Γεωργία και με την προσωπία πριν από δύο εβδομάδες από το γραφείο μου πήγε στην Μόσχα και συζήτησε μαζί του την υπόθεση της Γεωργίας και είπα θα έλεγα ναι ότι στην αρχή της θητείας μου υπήρχε εχθρό αλλά ακόμα μετά την παραπομπή του Νταρφούρ ε, άλλαξε τα πράγματα και ο πρόεδρος Μπούς ήταν σαφή υποστηρικτή των δυστηριοτήτων δικαστηρίου στην περίπτωση του Νταρφούρ και τα πιο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ζήτημα για τη ΣΥΠΑ ήταν ότι ο εισαγγελέα έχει ανεξαρτησία για να ασκήσει δίωξη. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησα την εξαρτησία αυτή για να ασκήσω δίωξη στην Κένια. Και πήταν θέση τον είπα, Πλήρη υποστήριξη, ανοιχτή υποστήριξη, δημόσια υποστήριξη. Πιστεύω ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Δεν θα υπογράψουν αύριο τη συνθήκη, εντάξει. Αλλά συνεργάζονται μαζί μα. Για αυτή τη ενία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξακολουθεί να ηγείται. Διότι περί αυτού πρόκειται. Καμιά φορά οι Αμερικανοί λένε, εάν δεν ηγούνται, τίποτα δεν συμβαίνει. Καλώ, σε αυτή την περίπτωση δεν ηγούνται και αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα, έχουμε πολλά παράδοξα εδώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κυρία Βερζιά. Χαίρομαι που παρευρίσκεστε εδώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Εγώ ήμουν μεταξύ όσων ε, είδαν ε, τη γέννηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με πολύ μεγάλη χαρά γιατί πραγματικά πρόκειται για μεγάλη πρόοδο για το διεθνές ε, δίκαιο. Και πραγματικά λυπούμαστε που κάποια μεγάλα κράτη δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη Σύμβαση της Ρώμης. Φαίνεται ότι κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον κάποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάποια δυσκολία να δεσμευτεί πλήρως με την Σύμβαση της Ρώμης, λόγω της ευθυγράμμισης ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καθώς ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διατηρήσουν την αντιμορισία για τους δικούς τους υπηκόους. Πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να καταδικάζει τέτοια γεγονότα. Εξάλλου, όπως είπατε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει τον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των μερών θα πρέπει να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία μια σειρά διατάξεων. Θέλαμε να μας πείτε αν αυτό έχει γίνει στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει ένα λόγο και μία δράση συνεπή επί όλων αυτών των θεμάτων. Και σας υποστηρίζω όταν λέτε ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη στα κράτη αυτά, προκειμένου να διασφαλίζουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε προκειμένου να εφαρμόζεται ο νόμος με πάσα αυστηρότητα. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με την έρευνα σε ό,τι αφορά τη Γουινέα. Ε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πως ε, εσείς ε, και η Νότια Αμερική και οι Αφρικανοί θέλουν να ξεκινήσουν ένα νέο σύστημα που θα έχουμε νέα προστασία των πολιτών από τα δικαστήρια, τα εθνικά και αν δεν γίνεται αυτό θα παρεμβαίνει το δικαστήριο και οι πολίτε χωρών που δεν είναι στο σύστημα δεν έχουν την ίδια προστασία. Έρχονται σε μένα άνθρωποι από τη Σρι Λάνκα, Λίβανο, Βυρμανία και μου ζητάνε παρέμβαση. Ε, λυπούμε, δεν μπορώ. Ε, δεν, δεν είναι οι χώρε σα μέλη και δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε από αυτή την έννοια έχουν λιγότερα δικαιώματα. Οπότε το σύστημα είναι ένα νέο σύστημα. Δεν το έχουν υπογράψει όλε οι χώρε του κόσμου, γύρω σε 130. Αλλά αυτοί προστατεύονται καλύτερα οι πολίτε του. Υπ' αυτή την έννοια ο ρόλος της Ένωσης ε, που παίζει ηγετικό ρόλο έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό επιμένω το πώς θα, ορίσουμε, πώς θα ορίσετε την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, γιατί μετά αυτό έχει σημασία για όλο τον κόσμο. Αλλά ακόμα και τρίτα μέρη που διαπράττουν εγκλήματα στα 110 αυτά κράτη μπορούν να διωχθούν. η Κωνσταντίνα, γιατί ήταν τόσο, τόσο δραστήρια στον Ταρφούρ και το εξήγησε γιατί ήμασταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας τόσο ισχυρής. Κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν έχουμε στρατό, οπότε ο νόμος μόνο μας προστατεύει. Οπότε μια χώρα η οποία δέχεται εισβολή πρέπει να προστατευτεί. Και λένε, εμείς πρέπει να παίξουμε ηγετικό ρόλο γιατί είμαστε μεγαλύτεροι από τις 26 χώρες στον κόσμο που δεν έχουν στρατό. Ε, εσείς είστε λίγο μεγαλύτερα από την Κωνσταντίνα, αλλά βλέπετε το, το σκεπτικό. Είναι σταθερή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε προνομιακή θέση. Δεν φαντάζεστε καν τέτοια σύγκρουση στην Ευρώπη. Έχετε και έναν περιφερειακό οργανισμό πάρα πολύ ισχυρό, οπότε βοηθάτε άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο τυχερές να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Και τα μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ευχαριστώ. Ντέβα. Um, Ευχαριστώ. Ίσως είναι κάπως λεπτό αυτό το θέμα, αλλά άκουσα ότι όταν ασκούνται διώξεις για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από πρώην ηγέτες ε, που έχει τιμωρησίας, ότι όλη η διαδικασία της ε, έρευνας κύλησε ομαλά αλλά τελικά θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί αν ε, κρίνονταν ενοχή δεν θα μπορούσαν να μπουν στη φυλακή. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να περιορίσουμε την ελευθερία αυτών των ανθρώπων. αν θέλετε, το οικονομικό άχθος θα πρέπει να το αναλάβουν και τα 27 κράτη-μέλη με ένα πλέον ε, δίκαιο τρόπο. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω αυτό. Δεν ε, είναι δίκαιο αρμοδιότητα αυτό το θέμα. Τα άτομα, οι οικογένειες των ατόμων που έχουν ε, καταδικαστεί θα πρέπει να βρίσκονται κοντά ε, έτσι λοιπόν ε, η καλύτερη ιδέα πάντοτε είναι ε, το άτομο να φυλακίζεται εκεί όπου βρίσκεται η οικογένεια του, τέλος πάντων είναι κοντά στην οικογένεια του. Όμως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό το θέμα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Να ευχαριστώ κύριε Οκάμπο, λέει κυρία Χαουτέλα. Τα σχόλιά σας ήταν πολύ ενδιαφέροντα για το πώς ε, χώρες ε, που δεν είναι συμβαλόμενα μέρη της συνθήκης τρέφονται στο δικαστήριο, όπως έγινε στην περίπτωση της Ρωσίας με την υπόθεση της Γεωργίας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο έγκλημα της ε, επίθεσης, αγκρέσιων. Πώς αυτό θα συμπεριληφθεί στο έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το σχολείο σας που λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα τώρα να ασκήσει μια πιο συνεπή εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και σε όλες τις εξωτερικές μας σχέσεις να βάλουμε και τη συνιστόσα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και φυσικά το Κοινοβούλιο μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε να προβάλλει περισσότερο το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μπορεί να εκπλήσει κάποιος το ότι ε, μπορείτε να έχετε, παραδείγματο χάρη, ακροατήριο ε, στη δί, στις δίκες στο δικαστηριό σας, ε, γιατί δεν προβαίνετε και σε web stream έτσι ώστε όλοι στον πλανήτη να μπορούν να παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου τη δίκη και να ξέρουν πώς δρά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κοιτάξτε, για το θέμα της επίθεσης, ε, εγώ θα εφαρμόσω ό,τι αποφασίσετε. Δεν ε, υιοθετώ εγώ την ομοθεσία. Τώρα για τις ακροάσεις, ε, συνήθως υπάρχει web streaming, όμως πολλές φορές για λόγους ασφαλείας πρέπει να διακόψουμε την αναμετάδοση. Όμως για το θέμα της εξωτερικής ε, διάσταση των εξωτερικών σχέσεων θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή χρονική στιγμή να συζητηθεί το θέμα αυτό. Πρέπει εσείς να κατανοήσετε το εξή. Ε, ρωτούν μερικοί γιατί είστε στην Αφρική ή ε, η Ευρώπη είχε πριν 60 χρόνια σειράξει, ενώ η Αφρική τι έχει σήμερα. Και εμεί του βοηθούμε να απειλήσουν τι σειράξει. Γιατί αν δείτε τι γίνεται στην Αφρική, υπάρχουν ε, τρία, ε, συγγνώμη, 30 κράτη τη Αφρική που είναι ε, μέλη, ενώ τα 26 τη Αφρική Ένωση δεν είναι τμήμα του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια ομάδα χωρών που προσπαθούν να αλλάξουν, αλλά έχουμε και μια άλλη ομάδα χωρών όπου συνεχίζουν να γίνονται εγκλήματα ε, από όσους έχουν την εξουσία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έτσι λοιπόν ε, δεν ε, πρέπει ε, να λαμβάνετε υπόψη τα σχόλια του πρόεδρου Μπασίλου χάρη του Κατάφη γιατί δεν είναι μέλη στην Κένια, λόγου χάρη, είναι σαφές ότι μας χρειάζονται για να ε, προλάβουμε εγκλήματα για το 2012, όχι μόνο στην Κένια και στην Τανζανία, ε, γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση, ε, γιατί αν καταρρεύσει το 2012 η Κένια, θα καταρρεύσει και η Τανζανία, γιατί θα καταρρεύσει η οικονομία και θα υπάρχουν και προβλήματα μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν ε, κοιτάξτε, μπορεί να είναι θέματα που πρέπει να τα διχειρίζεστε στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά στην Αφρική αυτά τα θέματα αφορούν την επιβίωση. Έχουμε τη βούληση 30 κρατών στην Αφρική που θέλουν να αλλάξουν και αυτά πρέπει να υποστηρίζει η Ευρώπη. Τρεις μέρες αφού ο Κατάφη έλεγε την απόφαση να μην συνεργαστεί με το δικαστήριο, Τρει μέρε μετά εγώ ήμουν ε, ε στο Ιναέδρα τη Αφρικανικής Ένωση, συναντήθηκα με τον ε, πρόεδρο Μπέγκη και κατέστη πολύ σαφές το τι συμβαίνει στην Αφρική. Θέλει η Αφρική ε, να αλλάξει. Υπάρχουν κάποιοι ηγέτε που προσπαθούν να αλλάξουν, όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που προσπαθούν να μην αλλάξει η κατάσταση στην Αφρική. Ευχαριστώ. Um, Κυρία Λούνατσεκ, να αναφερθώ σε κάτι που είπε και ο κύριος Λοχμπίλερ. Από ό,τι κατάλαβα τώρα υπάρχει ένα ταμείο για τα θύματα στο οποίο πρέπει να συνεισφέρουν ε, ε, συμβαλόμενα μέρη. Μπορείτε να μας πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το χρηματοδοτεί. Το χρηματοδοτεί τι κάνει. Για να δώσουμε κίνδυνο και στους άλλους. Υπάρχουν λεφτά ήδη. Τι γίνεται. Κάτι άλλο για τους εθνικούς συνδέσμους. Ε, δεν και μπορεί να το είπατε, ήρθα και λίγο αργά. Πάνω από 40 χώρες, είπατε, δεν έχουν ορίσει ήδη μόνιμο σύνδεσμο. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω, ε, αν υπάρχει πρόοδος.